okay, Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορώ να φωνάξω και πιο δυνατά αν δεν με ακούτε. Θα μπορούσατε να σταματήσετε τα πηγαδάκια και να καθίσετε στις θέσεις σας και να ξεκινήσουμε την ακρόαση. και ε, ίσως οι κάποιες από τις φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές να αποχωρήσουν γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Καθίστε παρακαλώ το ταχύτερο δυνατό γιατί θα έχουμε πρόβλημα χρόνου. Καθυστερήσουμε 10-15 λεπτά. Θα σας πω εκ των προτέρων ότι θα ξεπεράσουμε το χρόνο μας κατά 10 με 15 λεπτά. Δεν πρέπει να το να θεωρηθεί ότι φταίει η δική μας επιτροπή. Χαιρετίζω λοιπόν τον υποψήφιο επίτροπο, τον κύριο Αλμούνια, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους μας. Θα σας υπενθυμίσω ότι ο υποψήφιος επίτροπος έχει ήδη απαντήσει γραπτά το ερωτηματολόγιο το οποίο του έχει υποβληθεί και έχουν διανεμηθεί οι απαντήσεις του, οι στους βουλευτές σε όλες τις γλώσσες. Η αξιολόγηση θα γίνει από τη βάση της γενικής ικανότητος του Επιτρόπου, της προσήλωσής του στα ευρωπαϊκά θέματα, την ειδική γνώση για τα θέματα τα οποία είναι στην αρμοδιότητά του και την ικανότητα επικοινωνίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να είσαστε λίγο πιο γαλήνοι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Θα γίνουν με την γνωστή διαδικασία θα γίνει η ακρόαση αυτή, δηλαδή θα υπάρξει μια εισαγωγική παρέμβαση που δεν θα ξεπεράσει τα 10 λεπτά από τον υποψήφιο επίτροπο. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις των μελών, ξεκινώντας με ένα μέλος από κάθε πολιτική ομάδα. Στη συνέχεια, μετά από τον πρώτο γύρο ερωτήσεων από τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, θα υπάρξουν δύο ερωτήματα από την Επιτροπή Μεταφορών Αυτό γίνεται για να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους χωρίς να παρακαθίσουν σε όλη τη συνεδρίαση και θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Σας υπενθυμίζω ότι έχετε ένα λεπτό μονάχα για τις ερωτήσεις, δύο λεπτά για την απάντηση του υποψηφίου επιτρόπου. Δεν επιτρέπονται πολλαπλές ερωτήσεις. Ένα ερώτημα για τι ερωτη... για τις ερωτήσεις συνέχειας που πρέπει να, τις διπλωματικές ερωτήσεις που δεν θα πρέπει να εισάγουν νέα θέματα, θα πρέπει να είναι πάνω στα προηγούμενα θέματα και θα έχει μόνο ένα λεπτό να απαντήσει στις διπλωματικές ερωτήσεις ο υποψήφιος επίτροπος και επιφυλάσσουμε το δικαιώματος να ε, μην επιτρέψω ορισμένε ερωτήσει, εάν θεωρείς ότι είναι εκτό θέματο. <clears throat> Σα ζητώ επίση να μην μιλάτε πολύ γρήγορα και προτού δώσω το λόγο στον υποψήφιο επίτροπο, θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει ω προεδρεύουσα. Πρώτα απ' όλα, κύριε Αλμούνια, η Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων εκτιμά ιδιαίτερα την διαθεσιμότητά σας, όπως φάνηκε από τις απαντήσεις σας, να εργαστείτε σε ένα πνεύμα ανοιχτό και πνεύμα διαφάνειας με την Επιτροπή μας. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία να υπάρχει σωστή πληροφόρηση και έγκαιρη διαβίβαση νομοθετικών και μη νομοθετικών εγγράφων στο Κοινοβούλιο το ταχύτερο δυνατό, ακόμα και σε μορφή πρωτόλια, για να υπάρχει η δυνατότητα να λειτουργεί σωστά η διαδικασία λήψης αποφάσεων και ιδανικά αυτό θα πρέπει να ισχύει όχι μονάχα για αυτά τα οποία ζητούμε, αλλά και για πράγματα τα οποία γνωρίζετε εσείς ότι είναι πολύ πιθανό να μας ενδιαφέρουν. Θα εκτιμήσουμε λοιπόν ιδιαίτερα την δέσμευσή σας για αυτό το σημείο. Όπως ξέρετε, κατά τη διάρκεια της ε, χρηματοοικονομικής κρίσης, οι τρεις επιτροπές οι οποίες είναι αρμόδιες για τα θέματα αυτά, για τον ανταγωνισμό, της, ε, τα χρηματοοικονομικά <clears throat> και την ε, εσωτερική αγορά, συνεργάστηκαν μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή έχει ευθύνη για όλους αυτούς τους τομείς πολιτικής και εμεί θέλουμε να συμμετάσχουμε και να παίξουμε σημαντικό ρόλο στις πολιτικές αυτές. Επομένως, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δώσετε τον πρέποντα ρόλο στην Επιτροπή μας στους τομείς αυτούς. Στη γραπτή σας απάντηση είπατε επίσης ότι το θεσμικό σύστημα λήψης απόφασης της Κομισιόν για τον ανταγωνισμό είναι ένα ισχυρό σύστημα με εγγυήσει για την σωστή διαδικασία την δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα. Πολλές φορές όμως το σύστημα αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αναγνώσιμο και είναι δύσκολο να εξασφαλίσει κανείς ότι πράγματι όλες αυτές οι εγγυήσει τηρούνται και αυτό να μπορεί να το διακριβώσει κανείς εγκαίρος. Είχαν δυσκολίες λοιπόν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαπιστώσουν ότι πράγματι ισχύουν αυτέ οι εγγύησει. Είναι δύσκολο λοιπόν να έχουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο από τη δική μα πλευρά και ορισμένε φορέ ζητούμε περισσότερο από απλέ δηλώσει χωρί αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με αυτή τη διαδικασία. Ίσως στην τελική σα παρέμβαση στο τέλο θα μπορέσετε να μου δώσετε κάποια απάντηση σε αυτέ τι παρατηρήσει. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο στον υποψήφιο κύριο Επίτροπο. Ευχαριστώ. Thank you very much, Madam President. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, βουλευτές, τον Οκτώβριο του 2004, λίγο πάνω από πέντε χρόνια, βρέθηκα ενώπιον της ίδιας Επιτροπής και τότε μίλησα για τις ευρωπαϊστικές μου πεπιθήσεις και το γεγονός ότι θα ήθελα να συνεχίσω ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντολή που άρχισε τον Απρίλιο του 2004. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που τότε είπα. Τα τελευταία έξι χρόνια με ικανοποίησε ιδιαίτερα η συνεισφορά μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως η ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, η μετέπειτα ισχύς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ειρήνη και η σταθερότητα. Αυτός είναι ο απότερος στόχος και μια δημοκρατία και ελευθερία στην Ήπειρό μας καθώς και η τήρηση των κανόνων της αγοράς έτσι ώστε να είμαστε αποδοτικοί και δίκαιοι. Κατά, την, κατά το προηγούμενό μου χαρτοφυλάκιο και θητεία θεώρησα ότι πρέπει να έχουμε μια πιο ενωμένη Ευρώπη και πιο ενδυναμωμένη ως προς συνεργασία με τους εταίρους. Επίσης, θεωρώ ότι η Ευρώπη θα πρέπει να υπηρετεί του, τα 15 εκατομμύρια πολιτών που έχουν πληγεί από την πρόσφατη κρίση. Σε αυτή την περίοδο, μεταξύ το 2004 και την παρούσα στιγμή, προσπάθησα να είμαι συνεπής με αυτό το ιδεώδες και λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως το γράμμα των συνθήκων. Πολλές φορές ε, έγινε λόγος για την διαχείριση του χαρτοφυλακίου μου μέσα στα πλαίσια μιας καρποφόρας διαδικασίας κατά την άποψή μου. Κατά τη νέα περίοδο η στάση μου θα είναι η ίδια ως προς την αγαστή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για ε, πρόκριμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο έργο μας. Η κρίση άφησε πίσω πολλά θύματα, ιδιαίτερα νέους. Και εξαιτία της αρρωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, ισχύως των ε, συνθήκων μπορέσαμε να βοηθήσουμε όλα τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση, αυτή την πρόκληση με τα μέσα που διαθέτουν. Γι' αυτό χρειάζεται μια συντονισμένη έξοδος από την κρίση για να διασφαλίσουμε την ανάπτυξή μας και την ε, ανέλυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών. Η κρίση οδηγεί στην, στον επαναπροσδιορισμό της παγκόσμιας διακυβέρνησης έτσι ώστε να ενισχύσουμε την εξωτερική πτυχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πτυχή της εξωτερικής συνεργασίας. Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή φέρουμε μεγάλες ευθύνες κατά τα επόμενα έτη. Αναλαμβάνω αυτή την ε, ευθύνη με μεγάλη αισιοδοξία διότι θεωρώ ότι έχουμε τα κατάλληλα μέσα έτσι ώστε να ανταποκριθούμε επιτυχώς σε αυτές τις προκλήσεις. Και ιδιαίτερα με βάση μια νέα κοινοτική μέθοδο η οποία ενδυναμώθηκε με τη θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Στη, στο νέο χαρτοφυλάκιο θα αναλάβω συγκεκριμένες ευθύνες έτσι ώστε η Ευρώπη να βγει από την κρίση πιο ενισχυμένη, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην, ε, σε μια βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μαζί με την εσωτερική αγορά και το ευρώ πρέπει να διαδραματίσουμε συγκεκριμένο ρόλο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένα σημαντικό μέσο για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε σε παγκόσμια κλίμακα. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένοι όροι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται σε καλύτερη, σε καλύτερη θέση να ανταποκριθούν παγκοσμίως στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσουν και νέες θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει εδώ στην εσωτερική αγορά περισσότερο ανταγωνισμό και καλύτερη λειτουργία της αγοράς αλλά από πλευράς ε, των πολιτών, της προοπτικής των πολιτών που είναι και καταναλωτές, ο περισσότερος ανταγωνισμός σημαίνει περισσότερες επιλογές, καλύτερη ποιότητα, χαμηλότερες τιμές, καλύτερες υπηρεσίες και αυτό το έχουμε δει σε πληθώρα περιστάσεων. Θα καταβάλω κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να εφαρμόσω αυστηρά τους κανόνες ανταγωνισμού, έτσι ώστε να λάβω υπόψη και το αγγλοσαξονικό δίκαιο και να λάβω υπόψη και τις ε, νέες δυνατότητες ανταγωνισμού. Θα πρέπει να είμαστε αμερόληπτοι και να μην προωθήσουμε ιδιαίτερα συμφέροντα, ούτε να υπάρχει προτιμησιακή μεταχείριση ως προς συγκεκριμένους δικαιούχους. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα καρτέλ που είναι επιζήμια για τον ανταγωνισμό. Επίσης, προτείνω οι επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση να αποδυναμωθούν. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυστηρά το καθεστώς εποπτείας των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Και γι' αυτό θα πρέπει να μην δεχτούμε την δεσπόζουσα θέση ή τη δημιουργία δεσμος, δεσπόζουσας θέσης ορισμένων επιχειρήσεων. Δεν θα πρέπει λοιπόν να πληγεί ο ανταγωνισμός της, εξωτερικής, της εσωτερικής αγοράς. Πιστεύω ότι η παρούσα πλαισίωση ε, είναι διαφανής και ασφαλής έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, καταχρήσεις ως προς τον ανταγωνισμό. Βεβαίως μπορούν να επέλθουν βελτιώσεις, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα ε, φτάσουμε σε εγκάρσιες τομεακές ε, ε, αποφάσεις, ιδιαίτερα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ασφαλιστικών εταιριών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη συγκεκριμένες αποφάσεις εκεί όπου χρειάζεται και επίσης θα πρέπει να δούμε και τις οριζόντιες αποφάσεις και πού μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις ανακατηγορία. Ξέρετε ότι έχουν επέλθει πολλές βελτιώσεις. Θα πρέπει να βελτιώσουμε το εταιρικό ε, δίκαιο και να τηρηθούν οι αρχές ανταγωνισμού. Προτείνω να μελετήσω τις ε, διάφορες ε, προσεγγίσεις των συλλογικών συμβάσεων και συμφωνιών όπως ισχύει και σε άλλα μέρη του κόσμου. Επίσης θα λάβω υπόψη όλα τα σχόλια του Κοινοβουλίου πριν υποβάλω συγκεκριμένε προτάσεις έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει με βάση τη διαδικασία συναπόφασης ως προς τις κρατικές επιδοτήσεις θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς ανταποκρίνεται στη χρηματοπιστωτική κρίση. Τα κράτη-μέλη έχουν αναλάβει πολλές χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις με βάση τον τραπεζικό τομέα. Υπήρξε διευκόλυνση χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης χωρίς να υπάρξουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Τώρα θα πρέπει να έχουμε την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος έτσι ώστε μέσω και μακροπρόθεσμα να μπορέσει να, οδηγήσει, να οδηγηθεί στην χρηματοδότηση, σε χρηματοδοτήσεις χωρίς κρατικές επιδοτήσεις. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί βαθμία λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της οικονομίας και τους κινδύνους ως προς την οικονομική σταθερότητα. Πέρα από την υποστήριξη αυτή, οι κρατικές επιδοτήσεις θα πρέπει να δώσουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Η οικονομική κατάσταση, με βάση την οικονομική κατάσταση, η Επιτροπή θα πρέπει να κρίνει πότε θα πρέπει να επανέλθουμε στο προγενέστερο καθεστώς πριν από την κρίση. Και αν δεν αλλάξουν τα προσδοκόμενα, πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα ισχύσει στο τέλος του έτους. Η πολιτική αυτή θα οδηγήσει στην υπέρβαση της κρίσης, αλλά θα ήθελα να δούμε πώς να εξυγχρονίσουμε τον έλεγχο των δημόσιων επιδοτήσεων. Τα τελευταία χρόνια ορίσαμε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές ως προς την απασχόληση, το περιβάλλον και ούτω καθεξής και τώρα θα πρέπει να γίνει μια επαναξιολόγηση όλων αυτών των τομέων. Γενικότερα η πολιτική ανταγωνισμού θα ασχοληθεί με την επόμενη στρατηγική του 2020 και θα ορίσει τις ε, προτεραιότητες και τα μέσα έτσι ώστε να καταστήσουμε την οικονομία μας πιο δυναμική και πιο βιώσιμη. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να προωθήσουμε μια δυναμική και βιώσιμη οικονομία και έχουμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο. Η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να εγγυηθεί δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας κάτω από ε, δίκαιες και σωστές συνθήκες και να προωθήσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μέσα στα πλαίσια της ε, κοινωνικής συνοχής. Το πρωτόκολλο 26 και το άρθρο 104 της συνθήκης μας δίνουν τη δυνατότητα διακόπτη ο υποψήφιος διακόπτη για να επιβραδύνει λίγο το ρυθμό του, αλλά πρέπει τώρα να τελειώσει με την εισηγή. Λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να σας διακόψω, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, περνάμε τώρα στους βουλευτές από την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Γκάουζες, Πολ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχήν να σας, δεν τολμώ να πω να σας πω το καλό ήλθατε, γιατί σίγουρα σας γνωρίζουμε πολύ καλά στην Επιτροπή αυτή, αλλά ενώπιον της νέας Επιτροπής μετά τις ευρωεκλογέ. Θέλουμε να έχουμε από εσά σαφείς και δεσμευμένες απαντήσεις για τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Ως αρμόδιος για τον ανταγωνισμό γνωρίζετε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά δεν είναι αυτός σκοπός η πολιτική ανταγωνισμού σε οικονομικό επίπεδο. Η ρύθμιση του ανταγωνισμού και η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να έχουν σαν στόχο την ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να αρθεί το άχθος όταν είναι αδικαιολόγητο σε χρηματοοικονομικό επίπεδο των επιτροπών, των εταιριών, προ το όφελο των ίδιων των εταιριών και των καταναλωτών. Θέλω λοιπόν να σα ρωτήσω για δύο συγκεκριμένα θέματα τα οποία συζητεί αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο, το θέμα των συλλογικών αγωγών και επίση το θέμα των προστήμων σε περίπτωση παραβιάσεως του, των κανόνων ανταγωνισμού. Ξέρετε ότι πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμό 1 του 2003. Είσαστε έτοιμο να ακολουθήσετε την οδό του Κοινοβουλίου και να πάρετε ειδικά μέτρα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκοζέ. Σα ευχαριστώ για το ερώτημά σα. Σίγουρα η πολιτική του ανταγωνισμού δεν είναι αυτός σκοπό αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, ένα απαράγραπτο εργαλείο για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Σε σχέση τώρα με το συγκεκριμένο ερώτημά σας σε ό,τι αφορά τις συλλογικέ αγωγές, είναι πράγματι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να αποζημιώνουμε τα θύματα της κακής λειτουργίας των κανόνων του ανταγωνισμού. Δεν είναι το μόνο εργαλείο το οποίο χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε και σε άλλε περιπτώσει να αποζημιώνουμε του καταναλωτέ σε συλλογικό επίπεδο. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό πάντω είναι δύο πράγματα. Καταρχήν να δούμε ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο να συνδυάσουμε τι διαδικασίε για συλλογικέ αγωγέ σε περίπτωση ανταγωνισμού με συλλογικέ αγωγέ σε άλλε περιπτώσει για να μην δημιουργήσουμε μια διαδικαστική ασάφεια ή πολυσημεία. Και επίση <clears throat> να αποφύγουμε τις καταχρήσεις που παρουσιάζονται στις λεγόμενες class actions, στις συλλογικές αγωγές σε άλλες χώρες και εδώ υπήρξε προβληματισμός και από την Κομισιόν και από το Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο προβληματισμός και εγώ φυσικά βασίζομαι στην ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγώ προτιμώ αυτά τα θέματα να συζητηθούν μέσα στα πλαίσια της συναπόφασης. Ένα δεύτερο ερώτημα ήταν αυτό των των προστήμων. Τα πρόστιμα έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα για αυτούς οι οποίοι θέλουν να υπονομεύσουν τον ανταγωνισμό. Είναι λοιπόν ένα αποτρεπτικό εργαλείο το οποίο πρέπει να διατηρηθεί στο κατάλληλο επίπεδο. Αν δεν είναι αρκετά αποτρεπτικά τα πρόστιμα, οι επιχειρήσεις θα τα πληρώνουν και θα συνεχίζουν τις πρακτικές τους. Βάσει των αναλύσεων που γνωρίζω εγώ για τα θέματα αυτά, το επίπεδο αυτών των προστήμων είναι κατάλληλο αυτό το επίπεδο, σε γενικό επίπεδο, ώστε να υπάρχει αυτό το αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Γκοζές, πρέπει να επαναλάβω το ερώτημα για να μπορέσει να απαντήσει ο κύριος Επίτροπος. Υπάρχουν οι βόρειοι και οι νότιοι. Εγώ είμαι με τους νότιους και προτιμώ τις ε, εκτενείς απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Γκοζές, λέει ο κύριος Αλμούνια. Σας έλεγα ότι τα, κατά τη δική μου άποψη, κατά τις δικές μου αναλύσεις, έχουν ένα επίπεδο τα πρόστιμα που είναι συνεκτικό με τον αποτρεπτικό τους ρόλο, που είναι απολύτως απαραίτητο σε αυτή την πολιτική κυρώσεων. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν κυρώσεις ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή για τις εταιρείες ενός μονάχα προϊόντος ότι ο αντίκτυπος αυτών των προστήμων είναι πιο μεγάλος από ό,τι σε επιχειρήσεις που έχουν διαφοροποιημένη παραγωγή ή βρισκόνται μέσα σε ένα ευρύτερο οικονομικό όμιλο. Θα εξακολουθήσουμε να αναλύουμε αυτό το πρόβλημα. Μπορώ να σας πω όμως ότι τα πρόστιμα τα οποία έχουν αποφασιστεί από την Κομισιόν μετά από την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών του 2006 έχουν αποφασιστεί περίπου 50 επιβολές κυρώσεων έκτοτε αλλά μόνο σε τρεις περιπτώσεις το επίπεδο αυτών των προστήμων έφτασε το 10% που θεσπίζει ο κανονισμός ως το μέγιστο ποσό που μπορεί να φτάσει το πρόστιμο σε σχέση με τον κύκλο εργασιών μιας επιχείρησης. Um, Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στους σοσιαλιστές και δημοκράτες και στον κύριο Σάντσες Πρεζέδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να καλωσορίσω τον υποψήφιο επίτροπο κύριο Αλμούνια καλή χρονιά. Ελπίζουμε ότι θα είναι καλή και η πενταετία και όχι μονάχα το έτος το οποίο ακολουθεί. Δεν χρειαζόσαστε κάρτα ε, επισκεπτηρίου ενώπιον της Επιτροπής μας. Έχετε δείξει τα τελευταία χρόνια την ικανότητά σας για διάλογο και συνεργασίας με την Επιτροπή μας στα προηγούμενα καθήκοντά σας. Τώρα έχετε νέα καθήκοντα ως Επίτροπος Αρμοδιότητας και ως Αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή κρίσης και σε μια εποχή που ο ανταγωνισμός είναι πια παγκόσμιος όλο και περισσότερο, εγώ συμμερίζομαι αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος Τελόρ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ολοκλήρωσή της βασίζεται σε τρία στοιχεία. Τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων, τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών και την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών. Επομένως θα πρέπει να οδηγήσει ο ανταγωνισμός στα καλύτερα αποτελέσματα για να είναι προ όφελο των πολιτών και των καταναλωτών. Εγώ χαίρομαι για το ευρωπαϊκό πνεύμα το οποίο έχετε επιδείξει σε σχέση με την πολιτική ανταγωνισμού. Σε σχέση με τις ε, αγωγές θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα. μιλήσατε για τις καταχρήσεις στην περίπτωση των συλλογικών αγωγών, για την οριζόντια προσέγγιση. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι υπάρχει μια οριζόντια προσέγγιση που καλύπτει και όλα τα θέματα τα άλλα της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάντζες Πρεσέδο, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας επίσης. Προφανώς θα πρέπει να επαναλάβω ενώπιον της Επιτροπής σας ότι η στάση μου, όπως είπα στην αρχή, είναι μια στάση ανοιχτή για διάλογο και συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με όλους τους ενδιαφερόμενους. Θα εξακολουθώ να παραμένω σε αυτό το μήκο κύματο και θα προσπαθήσω να βελτιώσω αυτή τη διαδικασία τα επερχόμενα χρόνια. <clears throat> Συμφωνώ επίση για αυτό που είπατε για τη ρίση του Ζακ Τελόρ για το, λόγο, για το ρόλο του ανταγωνισμού και τη αλληλεγγύη σε ό,τι αφορά τι συλλογικέ αγωγέ. Όταν πρόκειται για συλλογικέ ζημίε που έχουν υποστεί οι καταναλωτέ, είπα προηγουμένω στην περίπτωση τη απάντηση στον κύριο Γκοζέ. Υπάρχουν οι αποζημιώσει λόγω σφαλμάτων επιχειρήσεων που δεν σέβονται τους κανόνες ανταγωνισμού, αλλά υπάρχει και περίπτωση αποζημίωσης για τοξικά ή ελλημα... ελαττωματικά προϊόντα. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν συντονισμός μεταξύ όλων αυτών των περιπτώσεων που είναι απαραίτητη μια συλλογική αποζημίωση η ελαττωματικα μπορεί να έλθει ενώπιον των δικαστηρίων. Θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε και κάποια εναρμόνιση των εθνικών διαδικασιών ενώπιον των δικαστηρίων και επίσης θα πρέπει να μπορούμε να εισαγάγουμε στο βαθμό του δυνατού μηχανισμούς οι οποίοι οδηγούν σε εξοδικαστική επίλυση αυτών των ε, προβλημάτων και παροχή αποζημίσεων για να μην υπάρξει υπερβολική προσφυγή στα δικαστήρια και να καταλήξουμε στις ε, υπερβολές των class actions που έχουμε δει σε άλλες χώρες. 30 ε, δευτερόλεπτα αν θέλετε να επανέλθετε. Όχι, ωραία περνάμε στους φιλελεύθερους και στην κυρία Γκουλάρ. Καλημέρα σας κύριε υποψήφι επίτροπε. Ε, είσαστε γνωστός και το έργο σας είναι γνωστό. Έχετε ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάχιο. Έχετε διευρυμένες ε, ευθύνες έτσι ώστε να καταπολεμήσετε τα καρτέλ, να βοηθήσετε τις ΜΜΕ, τους καταναλωτές, και πιστεύω ότι η πολιτική ανταγωνισμού στέφθηκε από επιτυχία στο παρελθόν. Υπάρχουν όμως πολλές αμφισβητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπήρξε υπερβολική απελευθέρωση της αγοράς. Μιλήσατε για πολίτες, καταναλωτές. Ίσως ο πολίτης δεν είναι μόνο καταναλωτής. Και αυτό θα πρέπει να σας απασχόλησει πώς θα επανισορροπήσετε την κατάσταση γιατί μας απασχολεί εμάς τους φιλελεύθερους ιδιαίτερα το θέμα πώς θα συμφιλιώσετε τους Ευρωπαίους με την πολιτική ανταγωνισμού. Ευχαριστώ την κυρία Γκουλάρ. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ευρωπαίος ε, πολίτης ε, είναι, αντιμάχεται μάλλον την ε, πολιτική υπέρ του καταναλωτή. Νομίζω ότι ε, θέλει να καταπολεμηθούν τα καρτέλ και επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση. Έχει αρνητική στάση ως προσεσμένες εθνικές επιδοτήσεις που στρεβλώνουν τον ε, ανταγωνισμό. Δεν θέλει προνόμια δηλαδή ο πολίτης ε, σε σχέση με την χορήγηση επιδοτήσεων ούτε στις επιχειρήσεις που μπορούν να καταχραστούν τις ε, ε, δεσπόζουσας θέσεις τους. Ακόμα και αν η διάσταση των επιχειρήσεων αποτελεί κάτι το θετικό στην πολιτική ανταγωνισμού γενικότερα. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις συνθήκες καταρχήν και τις διατάξεις που απορρέουν από τη συνθήκη. Οι συνθήκες η συνθήκη της Ρώμης αρχικά και όλες οι μεταγενέστερες ε, δημιούργησαν ένα παγκόσμιο πλαίσιο ανταγωνισμού. Θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο και επίσης θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την καλή λειτουργία της αγοράς. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από μια ρύθμιση της αγοράς που επιτρέπει την ύπαρξη ε, δημοσίων υπηρεσιών, κάτι το οποίο δεν μπορούν να παράσχουν οι αγορές από μόνες τους, να παρέχουν οι αγορές από μόνες τους και ποια είναι τα πλεονεκτήματα ε, βοήθειας ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι η πολιτική ανταγωνισμού, μάλλον είμαι υπέρμαχος της πολιτικής ανταγωνισμού στα πλαίσια της δική μου, μου θεώρησης και οράματος για την πολιτική ανταγωνισμού. Προέρχεστε από μία χώρα που ψήφισε υπέρ της συνθήκης, η δική μου όμως καταψήφισε τη συνθήκη. Θα ήθελα να σας επαναλάβω ότι θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά έτσι ώστε οι πολίτες να ταχθούν υπέρ των κρατικών επιδοτήσεων που να μην βλάπτει την εργασία τους. Πιστεύω ότι και τα κράτη-μέλη φέρνουν την ευθύνη, αλλά το δημόσιο χρήμα θα πρέπει να οδηγήσει σε επενδύσεις υπέρ του μέλλοντος, διότι πολλοί ε, δεν μπορούν να είναι υπόψη αυτά τα μακροοικονομικά δεδομένα. Συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να επεξηγήσουμε επακριβώς τα πλεονεκτήματα της πολιτικής ανταγωνισμού διαβάζοντας μόνο τη συνθήκη. Γι' αυτό ερμηνεύουμε τη συνθήκη, την επεξηγούμε και προβάλλουμε μια επιχειρηματολογία στη χώρα σας και σε πολλές άλλες χώρες θα καταβάλω κάθε προσπάθεια υπέρ μιας ε, δημοσιονομικής ε, πολιτικής με, την, ε, με μια συγκεκριμένη πειθαρχία. Πολλοί ακούν αυτά τα επιχειρήματα. Στο γαλλικό τύπο διάβασα για μια μελέτη η οποία αναφέρει ότι ο Γάλλος πολίτης ε, απασχολείται, μάλλον ανησυχεί ιδιαίτερα από το δημόσιο χρέος και επεξηγούμε τα πλεονεκτήματα της ε, καλής λειτουργίας της αγοράς. Δηλαδή να καταπολεμήσουμε τα καρτέλ, την ε, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, τη στρέβλωση ανταγωνισμού, έτσι ώστε να υπάρχει καλή χρήση των χρημάτων του φορολογούμενου. Τότε θα μας υποστηρίξουν. Αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε τη δημόσια διοίκηση έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει καλώς η αγορά. Συγγνώμη που σας σταματάω στο μέσο της ομιλίας. Ο κύριος Λάμπερτς από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και εμείς από την πλευρά των Πρασίνων έχουμε εκτιμήσει ιδιαίτερα μέχρι τώρα την ποιότητα του διαλόγου που έχετε διατηρήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι που τονίσατε ότι θέλετε και στα νέα σας καθήκοντα να συνεχίσετε να έχετε ένα διάλογο ποιότητος μαζί μας. Θέλω να σας εμπλέξω σε ένα θέμα που είναι κάπως δύσκολο, που μέχρι τώρα δεν έχει τύχει ίσως της πρέπουσας προσοχής από τις υπηρεσίες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάω για το δημοσιονομικό ανταγωνισμό. Μπορείτε να πείτε ότι δεν σας αφορά, αλλά είναι μια μορφή ανταγωνισμού που μπορεί να είναι αθέμητος και ιδίως μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά. Όταν ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγει στο νομικό του οπλοστάσιο ε, διατάξεις δημοσιονομικές που μοιάζουν με αυτές των φορολογικών παραδείσων και με τον τρόπο αυτό προσελκύει οι επιχειρήσεις και αποστερεί από τους γείτονές του φορολογικά έσοδα, αυτό οδηγεί σε μια στρέβλωση της αγοράς. Επομένω, αυτό που θέλουμε να ξέρουμε είναι ποια είναι η θέση σα σε σχέση με αυτό το πρόβλημα και ποιε είναι οι πρωτοβουλίε που θα λάβετε σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαμπέρ. Πρώτα απ' όλα η θέση μου και η θέση της τωρινής Κομισιόν και της επερχόμενης Κομισιόν είναι ότι είμαστε κατά των φορολογικών παραδείσων. Αγωνιζόμαστε εναντίον τους. Μέσα στο, τελικό, μέσα στο τελευταίο το διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια μετά από τους συνόδους των G20 και με πρωτοβουλίες της Κομισιόν, ο αγώνας κατά των ε, φορολογικών παραδείσων και κατά των κυβερνήσεων οι οποίες δεν συνεργάζονται μαζί μας έχει ενισχυθεί και ελπίζουμε ότι θα έχουν αποτελέσματα. Ξέρετε ότι υπάρχουν τέτοιες πολλές συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού χαρακτήρα μετά από τα πρώτα συμπεράσματα των G20. Δεν είναι εύκολα, πρέπει να συνεχίσουμε αυτό τον αγώνα. Τι γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τη φορολογία, σε επίπεδο ανταγωνισμού. Στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους δεν μπορεί να γίνει φορολογικός ανταγωνισμός μέσω επιλεκτικών φόρων. Αλλά μεταξύ ενός κράτους και άλλους κράτους, οι συνθήκες και η πάγια νομολογία μας λέει ότι είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας η θέσπιση του επίπεδου φορολογίας βάσει των οδηγιών και των κανονισμών που ισχύουν για το ΦΠΑ κτλ. Ίσως εσείς και εγώ θα θέλαμε να υπάρξει ένα διαφορετικό πλαίσιο συνεργασίας σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Αλλά ω Επίτροπο Ανταγωνισμού, εγώ δεν μπορώ παρά να σεβαστώ τι συνθήκε. Το κατανοείτε. Το κατανοείτε. Να μια σαφή και αναγνώσιμη απάντηση. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ευρωπαίο πολίτη και όπω έλεγε η Σιλβί Γκουλάρ, αν θέλουμε αυτή η Ένωση να φαίνεται ότι είναι πραγματικά μια Ένωση ενώπιον των πολιτών, θα πρέπει να δείξει ενδιαφέρον η Ευρωπαϊκή Ένωση και να επανέλθει στα θέματα αυτά των συνθηκών και της ε, νομολογίας, γιατί αλλιώς ο πολίτης θα έχει την εντύπωση ότι και πάλι γίνεται προς το συμφέρον ορισμένων επιχειρήσεων που αποστερούμε ε, κονδύλια από τις δημόσιες υπηρεσίες. Θα δούμε τι ακριβώς λέει η νομολογία για τα θέματα αυτά, αλλά εμείς δεν μπορούμε να υπαγορεύσουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Νομίζω όμως ότι μπορώ μέσα στις ε, αντιδράσει πολλών κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην κρίση στην χρηματοοικονομική, μπορώ να διακρίνω εκεί μια κοινή θέση έναντι τη φορολογία που είναι μια αλλαγή σε σχέση με την ε, κυρίαρχη κουλτούρα τη δεκαετία του 1980-1990. Νομίζω ότι αρχίζει να υπάρχει μια κίνηση από τα κράτη-μέλη και θα επανέλθουμε στη συζήτηση του θέματος αυτού, ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ. Η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και να σας ευχαριστήσω εκ μέρους ομάδας μου για την ε, συνεισφορά σας. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ ε, στις κρατικές ενισχύσεις και στα προσωρινά αυτά μέτρα, ιδιαίτερα όσον αφορά της, ε, τη χρηματοδότηση σε εταιρείε σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και μετά από αυτά τα μέτρα αποφάσισε η σχετική Γενική Διεύθυνση να παρέμβει για να υπάρξει μια φυσιολογική απόσυρση αυτών των μέτρων. Μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας καθώς ε, και πώς θα διασφαλιστεί ότι η άποψη της ε, κοινή γνώμης είναι μια άποψη που ε, αφορά την, που κλείνει προς την ε, αντικειμενικότητα και την δικαιοσύνη. Πώς ε, σκοπεύετε λοιπόν να διασφαλίσετε αυτή την δικαιοσύνη, την διαφάνεια και τέλος αν σκοπεύετε να παίξετε ένα ρόλο εποπτείας των εταιριών αυτών οι οποίες δέχτηκαν αυτές τις παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ. Όπως ξέρετε η Επιτροπή υιοθέτησε τέσσερις ε, ανακοινώσεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις κρατικές ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης. Μια γενική ανακοίνωση για τον τραπεζικό τομέα, μια άλλη για την ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου και άλλη μια για τις εγγυήσεις ε, και για τα στοιχεία ενεργητικού. Νομίζω όλα αυτά τα στοιχεία έχουν συζητηθεί και εντός Κομισιών και Εντό του Κοινοβουλίου και είμαι σίγουρος πως θα ξέρετε πως οι συζητήσεις που είχαμε στην ε, προηγούμενη θητεία ήταν και με το ΕΚΟΦΗΝ με τα κρατη οπότε υπήρχε ένα πλαίσιο για να υπάρχει μια συνοχή για ε, δύο ίδια αποφάσεων που αναγκαστήκαμε να ευθύσουμε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Δηλαδή πρώτον να δώσουμε έγκριση ή όχι στα σχέδια που εγκρίθηκαν σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη-μέλη, από πολλά κράτη-μέλη, για να στηρίξουν το τραπεζικό σύστημα, το χρηματοπιστωτικό τομέα και προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές για να υπάρχει η συμμεταχείριση των διαφόρων σχεδίων που δεν ήταν βέβαια τα ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη και δεύτερον τη μεταχείριση της κάθε μεμονωμένης περίπτωσης πρώτα απ' όλα των τραπεζών που διασώθηκαν που είχαμε ξεκινήσει το 2007 με τις πρώτες τέτοιες περιπτώσεις και μετά με τις τράπεζες που για τον χύψη λόγο είχαν λάβει κρατικές ενισχύσεις. Τώρα αποφασίζουμε τι συνέχεια θα δοθεί σε αυτά τα προγράμματα και λαμβάνουμε αποφασικά τα περίπτωση. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, παρατείνονται τα εθνικά σχέδια αυτά γιατί υπάρχουν ακόμη σαφείς κινδυνοί για τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σε άλλες περιπτώσεις ε, αναλύοντας τα σχέδια αυτά αναδιάρθρωσης ε, ανάλογα με το κάθε τράπεζα. Νομίζω πως κάνουμε καλή δουλειά και θα συνεχίσουμε γιατί πολλές αποφάσεις θα πρέπει να υιοθετηθούν τους ερχόμενους μήνες και το επόμενο έτος και ταυτόχρονα συζητάμε μεταξύ μας με το ΕΚΟΦΗΝ και με το Κοινοβούλιο πότε και διακόπτη πρόεδρος τον κύριο Αλμούνια. Με συγχωρείτε, θέλετε να επανέλθετε. Ναι, βεβαίως. Ξέρω πως ε, με το προηγούμενο χαρτοφυλάκιό σας ε, είχατε κάποια αίσθηση για το ποια χρηματοπιστοποιητικά ιδρύματα θα μας ε, ανισχύσουν. Μπορείτε να μας πείτε Τώρα τι θα γίνει στην πλευρά του ανταγωνισμού. Αυτό το οποίο με ενισχύει και στην προηγούμενη μου δουλειά και σε αυτή είναι πρώτα απ' όλα να αποφύγουμε τον περισσότερο, τον περαιτέρω κίνδυνο, δηλαδή να μην ενθαρρύνουμε όσους είχαν κακές αποδόσεις να ακολουθήσουν την πορεία που ακολουθούσαν και να συνεχίσουν να λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις. Δεύτερον, για να υπάρξει δίκαιος ανταγωνισμός, να διασφαλίσουμε πως ε, τα επιχειρηματικά μοντέλα αυτών των ε, τραπεζών είναι βιώσιμα έτσι ώστε να συνεχίσουν να δανείζουν στην πραγματική οικονομία. Αυτός είναι ο ρόλος του τραπεζικού τομέα. Και βεβαίως να μην αδικήσουμε όσους τα πήγαν καλά, που δικαίως βεβαίως ζητούν από την Κομισιόν μας λένε μην επιτρέψετε σε αυτούς που δεν θα επιβίωναν από μόνοι τους ε, να βγουν καλύτερα από μας. Οπότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί παραδείγματος χάρη είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θυμάμαι την τελευταία συζήτηση του ΕΚΟΦΗΝ, είχε πει η Νέλη Κρούς, ε, η προκάτοχός μου, παρακαλώ να είστε σόφρονες γιατί κινδυνεύει εδώ πέρα η δημοσιονομική σταθερότητα. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην Κούε τώρα και στον κύριο Κλούτε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αλμούνια, έχω κάποια ερωτήματα και εγώ για τις ε, τράπεζες. Είμαι από ένα κράτος μέλος ε, στο οποίο πέρα από τις ιδιωτικές τράπεζες υπάρχουν και οι τράπεζες των κρατηδιών και τα ταμιευτήρια που είναι πάρα πολύ ίσχυρα, τα οποία δέχτηκαν πάλι επίθεση από την Κομισιόν. Εσείς, ε, η Κομισιόν τα θεωρεί στρεβλωτικά του ανταγωνισμού, αλλά από την άλλη τα ταμιευτήρια αποδείχτηκαν πως αντέχουν στην κρίση, οπότε νομίζω πως ε, έχουμε ένα λογικό τραπεζικό σύστημα. Η άποψή σας ως ε, Υποψήφιο επιτρόπος ανταγωνισμού, ποια είναι για, τις, για το σύστημα αυτό των δημόσιων τραπεζών. Και εγώ, και εγώ προέρχομαι από μια χώρα η οποία έχει πολλές ιδιωτικές τράπεζες και ιδιαίτερα τράπεζες αποταμιεύσεων και επίσης τράπεζες που λειτουργούν συνεταιριστικά. Ε, είμαι υπέρμαχος τους ε, γεγονότος ότι οι χρηματοπιστωτικές αυτές οντότητες είναι καλές ή κακές ανάλογα με το πώς τις ε, διαχειριζόμαστε, δηλαδή κατά πόσο είναι φερέγγιες σε σχέση με την πιστοδοτική τους ικανότητα και να μην οδηγούν σε κινδύνους που μετά θα πρέπει να πληρώσουμε όλοι οι φορολογούμενοι από την τσέπη μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι έτσι θα πρέπει να ανταποκριθώ ως Επίτροπος Επιθεμάτων Ανταγωνισμού. Mm, ε, ναι. Κοιτάξτε βεβαίως το ισχυρό του σημείο ήταν ε, ε, μέχρι τώρα το ότι ήταν δημόσιες τράπεζες και είχαν την εγγύηση του, του κράτους και έκαναν πολιτική, δηλαδή ενίσχυαν ειδικά στη Γερμανία τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς τα τελευταία χρόνια μεγάλες τράπεζες δεν άνοιγαν λογαριασμούς για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Ε, και εξαρτήθηκαν αυτές από αυτή τη δομή στην οποία ασκείται κριτική. Οπότε εγώ ερμηνεύω την απάντησή σας, πείτε μου αν κάνω λάθος, ότι θα συνεχίσετε να επιτίθεστε στην μορφή αυτή που έχουν οι δημόσιες τράπεζες στη Γερμανία. Ε, Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων μου θα κρατήσω τις διαδικασίες ανταγωνισμού όπως έκανε και ο Μισελ Μπαρνιέ ως προς τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε να δούμε το θέμα της δημοσιονομικής ρύθμισης και των εποπτικών αρχών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να τηρούνται αυτές οι προδιαγραφές. Και αυτό αφορά ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Είχαμε πολύ καλά παραδείγματα διαχείρισης κατά τη διάρκεια της κρίσης από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δεν έχουν τη μορφή της τράπεζας, αλλά λειτουργούσαν ως ταμιευτήρια, για παράδειγμα, και ε, πολλούς οργανισμούς όπου υπήρχαν, υπήρξε κακοδιαχείριση ή έγιναν κακές επενδύσεις από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς δηλαδή. Ε, υπήρχαν επενδυτικοί οργανισμοί, ασφαλιστικοί οργανισμοί που γνωρίζουμε πολύ καλά όπως τις είπα που δεν διαχειριστήκαν καλά το ολοπλαίσιο. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην είμαστε ε, θύματα της κρίσης και ε, σε αυτό ευθύνεται η καλή διαχείριση και η καλή εποπτεία. Περνάμε τώρα στον κύριο Μπλουμ. Με συγχωρείτε που εγώ θα αναφερθώ σε κάποια διαφορετικά ζητήματα. Με εντυπωσίασαν κάπως οι Βρετανοί συνάδελφοι. Νομίζω πως είχαμε το λάθος άτομο εδώ πέρα. Μετά αν θέλω να ξεκαθαρίσω ένα ζήτημα. Είσαστε μέλος της μαρξιστικής στέριγας του Σοσιαλιστικού Κόμματος ε, της Ισπανίας ήσασταν ε, μέλος κυβέρνησης ε, της Ισπανίας το 86-91 και κατά της ανεξαρτησίας των βαλτικών κρατών και ήσασταν επίσης μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ήμουνα μέλος της ισπανικής κυβέρνησης του ΠΕΣΟΕ, στο οποίο ανήκω από το 1974, και η κυβέρνηση του ΠΕΣΟΕ, του Ισπανικού ε, Σοσιαλιστικού Κόμματος, αν μιλήσετε με τον επίτροπο, με τον, με τον ε, καγκελάριο Κολ, ήταν η χώρα αυτή που έχει υποστηρίξει από την αρχή την ενοποίηση της Γερμανίας και τη διαδικασία δημοκρατικοποίησης στις χώρες Κεντροανατολική Ευρώπη, που είναι σήμερα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή λοιπόν η διεύρυνση τη Ευρώπη υποστηρίχθηκε πάντα από το κόμμα μου και από μένα χωρί καμία απολύτω επιφύλαξη και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τι επερχόμενε διευθύνσει. Σε σχέση με τι ενδεχόμενε συμφωνίε ή συμπράξει πολιτικών κομμάτων μέσα στι βασικέ μα αρχέ σαν Ευρωπαίοι, που είμαστε ελεύθεροι και δημοκράτες, είναι ότι όλες οι ιδέες θα πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα και όσο εκφράζονται χωρίς βία είναι εξίσου έγκυρες και θεμητές είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Όχι, νομίζω ότι έχετε απαντήσει θαυμάσια το ερώτημά μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα προχωρούμε στον κύριο Μάρτιν για τους μη εγγεγραμμένους. Έχετε το λόγο κύριε Μάρτιν. Hans Peter Μάρτιν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, οπωσδήποτε είστε επαγγελματίας και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Εάν υπάρχει... εάν υπήρχε η δυνατότητα να αξιολογηθεί μεμονωμένα ο κάθε υποψήφιος, εσείς δεν θα είχατε καμία ανησυχία. Κάποιοι συνάδελφοι, ο κύριος Κάρας, παραδείγματος χάρη, λέει πως έχουμε τώρα τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά υπάρχουν τάσεις από πλευράς ε, Συμβουλίου με την υποστήριξη της ε, Κομισιόν να μην ε, έχει τα πλήρη δικαιώματα της συναπόφασής του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κάποια κόλπα θεωρείτε κι εσείς ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και τι σκοπεύετε να κάνετε για να εμποδίσετε κάτι τέτοιο, για να μπορέσει δηλαδή να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προφανώς ούτε προσωπικά, ούτε σαν μέλος της ε, προηγούμενης και της επερχόμενης Κομισιόν, εγώ δεν έχω δει καμία μορφή δισταγμού ή οποιαδήποτε προσπάθεια να περιοριστεί η εμβέλεια της συναπόφασης. Εγώ νιώθω πολύ ικανοποιημένο που η συνθήκη της Λισαβόνας διευρύνει ακόμα περισσότερο το χώρο της συναπόφασης. Είναι σημαντικός λοιπόν ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην ε, νομοθετική διαδικασία και στον τομέα αυτό που έχετε αναφέρει, στην πρωτοβουλία αυτή που δεν, υπάρχει που δεν υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες στον τομέα του ανταγωνισμού, αλλά αυτή που αναφέραμε προηγουμένως, που είναι αυτή για τις ε, συλλογικές αποζημιώσεις, έχω τονίσει ότι νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μέσω της διαδικασίας συναπόφασης που εμπλέκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, γνωρίζοντας όπως και εσείς, ότι αυτό βασίζεται στις νομικές βάσεις που μπορούμε να βρούμε για να θεσπίσουμε, για να διεκπαιρεώσουμε αυτά τα θέματα, γιατί υπάρχουν νομικές βάσεις οι οποίες δεν απαιτούν τη συναπόφαση. Έχετε συμπληρωματικό ερώτημα. Υπό το φως ε, των όσων είπατε, θα υποστηρίζατε παραδείγματο χάρη παρουσία βουλευτών στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Και βεβαίω ξυπακούτε πως μπορεί να είναι και εδώ παρόν ε, το Συμβούλιο. Αν ρωτάτε για τις σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν, εγώ σας λέω ότι θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ, πλαισίου μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν και έτσι θα ενισχύσουμε και θα βελτιώσουμε τον τρόπο της λειτουργίας των σχέσεών μας. Νομίζω ότι ήδη και στην προηγούμενη θητεία της Κομισιόν ήταν πολύ καλές αυτές οι σχέσεις από θεσμική έποψη. Σε, σχέση με τις, ε, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις σας με το Συμβούλιο, θα μου επιτρέψετε να παραπέμψω το θέμα αυτό στις αρχές του Συμβουλίου. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος για να ερμηνεύσω τη θέση του Συμβουλίου ή του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτό το σημαντικό ζήτημα. Okay, thank you very much. Um... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσουμε ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών γιατί έχετε στο χαρτοφυλακείο σας και ζητήματα μεταφορών. Πρώτα απ' όλα λοιπόν τον λόγο έχει ο κύριος Μαρινέσκου, δεν ξέρω που βρίσκεστε. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, από πρώτης ε, πρώτου 2010 απελευθερώθηκαν οι διεθνείς μεταφορές επιβατών, είχαν ήδη απελευθερωθεί οι μεταφορές φορτίου εμπορευμάτων και υπάρχουν ακόμα εταιρείες στην ιδιοκτησία των κρατών μελών που μεταφέρουν και επιβάτες και εμπορεύματα και υποφελούνται από τις κρατικές ενισχύσεις. Ταυτόχρονα οι μεταφορές είναι πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία για τους πολίτες της Ένωσης. Πώς βλέπετε το μέλλον Όσον αφορά το μελλοντικό σου χαρτοφυλάκιο, δηλαδή τον ανταγωνισμό και τις κρατικές ενισχύσεις. Όπως ε, γνωρίζετε, στην ε, νέα κατανομή καθήκοντων και χαρτοφυλακίων, ο πρόεδρος Μπαρόσο. πρότεινε να ασχοληθούμε και με το θέμα των εθνικών επιδοτήσεων μέσα στα πλαίσια της Γενικής Διεύθυνσης ε, Τρέν. Αυτές οι επιδοτήσεις, αυτές οι ενισχύσεις, σε αυτές τις ενισχύσεις ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ε, περιπτώσεις όπου θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τις κρατικές επιδοτήσεις στα πλαίσια των ΔΕΚΟ. Ε, υπάρχουν σαφή κριτήρια από πλευράς ε, νομολογίας, αλλά έχουμε να κάνουμε με μια νέα συνθήκη όπου στο άρθρο 14 που αφορά τις ε, δημόσιες μεταφορές και το άρθρο 106 που αναφέρεται στη νέα νομική βάση σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές γιατί μιλάμε για ένα quality framework, όπως όρισε ο πρόεδρος Μπαρόσο. Δεν είναι καθόλου απλό αυτό το ζήτημα. Ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών ε, συγκεντρώνονται πολλές ε, πτυχές αποφάσεων που δεν είναι καθόλου εύκολες. Δηλαδή, τι είναι δημόσια υπηρεσία και τι είναι η οικονομική δραστηριότητα στα πλαίσια του ανταγωνισμού, αλλά έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια μέσα στα πλαίσια τομέων που έχουν απελευθερωθεί και στο παρελθόν, όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές και μέρος των οδικών. Είπατε προηγουμένως ότι οι, δημόσιες, οι, μεταφορές, οι δημόσιες μεταφορές δίνουν μια σημαντική υπηρεσία στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να εξασφαλίσουμε την ελευθερία ανταγωνισμού και στην αγορά των μεταφορών. Βέβαια υπάρχουν και μονοπόλια σε ό,τι αφορά τις δημόσιες μεταφορές, παραδείγματος χάρη στην, περί, περίπτωση της ε, περιοχής του Παρισιού. Οι δημόσιες υπηρεσίες, το RER έχει και το RTP έχουν ένα μονοπόλιο. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι τέτοιου είδους μονοπόλια είναι δυνατά να υπάρχουν και πρέπει εδώ να τηρηθεί μια αρχή αμεβαιότητος, δηλαδή ότι αυτοί που έχουν ένα μονοπόλιο το οποίο ε, καλύπτεται από την κρατική υποστήριξη δεν θα πρέπει να είναι εκτός των ε, αγορών άλλων εταιριών σε άλλες χώρες. Όπως ξέρετε, μιλάμε πάντα για μια μορφή περιορισμού των ε, του πεδίου εφαρμογής των εταιριών κοινού, κοινοφελούς χαρακτήρα. Αυτό είναι κάτι που είναι στην εκτίμηση των κρατών μελών και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να κάνουμε ε, ενδελεχή εξέταση της κατάστασης και όχι να δημιουργούμε γενικές συλλήβδιν κατηγορίες. Θα πρέπει να δούμε τα θέματα αυτά σε όλη τη λεπτομέρειά τους. Εγώ προτιμώ να μην απαντήσω για αυτό το συγκεκριμένο θέμα το οποίο αναφέρετε. Καταγράφω αυτό το οποίο εσείς αναφέρατε καταγράφω το ενδιαφέρον σας για αυτό το θέμα, θα το αναλύσω αυτό το θέμα και σε κάποια μεταγενέστερη ευκαιρία ίσως θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε σε λεπτομέρεια. Δεν θέλω τώρα να προκαταλάβω μια θέση, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να αυτοσχεδιάζω σαν Επίτροπος Ανταγωνισμού χωρίς να ξέρω τις λεπτομέρειες όλων των στοιχείων που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση και ιδιαίτερα για τα νομικά ζητήματα τα οποία εμπλέκονται. Αυτό το κάνουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ, λέει ο κ. Ευχαριστώ λέγει η Πρόεδρος. Προχωρούμε τώρα στον κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι στην Επιτροπή Μεταφορών, Αντιπρόεδρος και θέλω να ρωτήσω τον νέο Επίτροπο για τις ε, κρατικές ε, ενισχύσεις στον τομέα των μεταφορών που πέρασαν στη δική σας Γενική Διεύθυνση ως αρμοδιότητα. Οπότε πώς θα συνεργαστείτε με τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών για να λάβετε υπόψη τον συγκεκριμένο τομέα των μεταφορών στις ε, κρατικές ενισχύσεις και πιο συγκεκριμένα με τους κανόνες κρατικής ενίσχυσης για τα λιμάνια. Η προηγούμενη Κομισιόν είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει γρήγορα να φέρει νέους ε, κανόνες το 2009 πέρασε το 2009 και το ερώτημα τελικά είναι πότε θα έρθει η νέα πρόταση για τις κρατικές ενισχύσεις των λιμανιών. Δεν είναι καθόλου απλό να μεταφέρονται ε, οι ευθύνε και τα καθήκοντα σε σχέση ε, με τις κρατικές ενισχύσεις από ένα χαρτοφυλάκιο σε ένα άλλο αλλά η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για αυτές τις κρατικές ανισχύσεις στη Γενική Διεύθυνση Τρεν θα πλαισιωθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Και ε, όλα αυτά εντάσσονται στις ε, μεταφορές. Άρα έχει μεγάλη σημασία ο συντονισμός ε, των επιτρόπων ανταγωνισμού και μεταφορών. Το ίδιο ισχύει και στη συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων όπως ε, μεταφορές και ανταγωνισμός. Ως προς το θέμα στο οποίο αναφερθήκατε τις ε, γενικές κατευθυντήριες γραμμές ε, για τους λιμένες, διενεργείται μία μελέτη, έχει αναλευθεί μία εργασία, θα φτάσουμε σε συμπεράσματα στους επόμενους μήνες και το θέμα εντάσσεται στις αρμοδιότητες ε, του χαρτοφυλακίου ανταγωνισμού μέσα στα πλαίσια των μεταφορών. Μία ακόμα ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε συγκεκριμένα πότε θα έρθει αυτή η πρόταση. Φέτος, πριν το καλοκαίρι. Και δεύτερο ερώτημα κάποια μέλη της Επιτροπής ε, Μεταφορών κοιτάνε τον ανταγωνισμό μεταξύ των μέσων ε, μεταφοράς. Κάποιες ε, πληρώνουν κάποιους φόρους, άλλοι όχι. Π.χ. η κυροζήνη είναι αφορολόγητη. Είναι μια πτυχή την οποία θα εξετάσατε τι θα κάνετε με τη διαφορά των φόρων που υπάρχουν στα διάφορα μέσα μεταφοράς ειδικά στο, ναι, στον τομέα των μεταφορών. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία για το πότε θα εισαχθούν αυτά τα μέτρα, διότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο υπόκειται σε αλλαγές. Αλλάζει δηλαδή το χαρτοφυλάκιο, υπεύθυνο χαρτοφυλακίου. Δηλαδή έχει σημασία για το πότε θα αναλάβει τα καθήκοντά της η νέα επιτροπή, το οποίο εξαρτάται από εσάς. Το θέμα ΦΠΑ δεν αφορά μόνο τον ανταγωνισμό, διότι μιλήσαμε και για φορολογικά πριν. Θα πρέπει να δούμε τις ε, επιχειρήσεις που θα πρέπει να τύχουν τις ίδιας μεταχείρισης που δεν νομίζω ότι πρόκειται για το ίδιο. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού. Είναι ένα θέμα πολιτικής μεταφορών που σχετίζεται με μια φορολογική πολιτική. Φορολογική πολιτική η οποία είναι πολύ δυσχερής, πολύ σημαντική αλλά και πολύ δύσκολη να επινοηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι υπόκειται σε ομοφωνία. Θα θυμόσαστε στο ΕΚΟΦΗΝ ε, ότι έγινε μια συζήτηση για το ΦΠΑ που θα έπρεπε να επιβληθεί για την κυροζήνη και θυμόσαστε πώς κατέληξε αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τα μέλη της Επιτροπής ε, Μεταφορών. Ξαναπερνάμε στα μέλη της Επιτροπής Συνομικών Θεμάτων και τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Γκαρθία Μαγκάλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε κύριε Υποψήφιε Επίτροπε. Όπως είπατε στην εισαγωγική σας παρέμβαση, καθ' όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης τα κράτη-μέλη χρειάστηκε να λάβουν μια σειρά από ετερογενή αλλά πολυδάπανα μέτρα για να διασώσουν ορισμένες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Τώρα όμως πρέπει εμείς να βγούμε από την κρίση το 2010 και στη συνέχεια θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Το πρώτο ερώτημα που έχω να σας θέσω είναι τι θα κάνετε εσείς ως Επίτροπος Ανταγωνισμού ώστε οι φορείς αυτοί οι πιστοτικοί οι οποίοι πήραν υποστήριξη από δημόσιο χρήμα δεν θα βρεθούν στο τέλος σε καλύτερη ανταγωνιστική θέση έναντι των επιχειρήσεων των τραπεζών που ήταν πιο σόφρονες και προσεκτικές. Και δεύτερον, τι μέτρα θα λάβετε ώστε οι τράπεζες να μην επανέλθουν στις τολμηρές με σε εισαγωγικά δράσεις που οδήγησαν στην κρίση και έχουμε μιλήσει πάντα για δημόσιες ε, ε, ενέργειες διασώσεως οι οποίες θα πρέπει όμως να είναι πιο προσεκτικές. Ευχαριστώ κύριε Μαργάιο. Καταρχήν, δεν ήταν όλες οι δημόσιες επιδοτήσεις για τον πιστοτικό τομέα, για τις χρηματοοικονομικές αυτές, ε, όλες αυτές που πήγαν σε αυτές τις επιχειρήσεις, μάλλον πήγανε όχι επειδή ήταν σε κατάσταση πτώχευση οι επιχειρήσεις αυτές, αλλά για να αποφύγουν να δημιουργηθεί κίνδυνος για την φερεγγιότητα αυτών των τραπεζών που μπορούσε να οδηγήσει σε γενικότερους συστημικούς κινδύνους για το χρηματοοικονομικό σύστημα και την ε, οικονομία συνολικά. Εγώ συμφωνώ μαζί σα ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατό να επανέλθουμε σε πραγματικές συνθήκες ανταγωνισμού, με ίσες συνθήκες ανταγωνισμού όλων των φορέων στην αγορά. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να ε, ζητήσουμε από αυτού οι οποίοι πήραν από επιδοτήσεις και βοήθειες στα σχέδια των ε, αναδιαθρώσεών του να γίνουν Βιώσιμε σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό τους μοντέλο σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο και να υπάρξουν επενδύσεις από τη δική τους πλευρά για να μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν την επιστροφή των αρρωγών και να εξασφαλίσουν τη σωστή κατανομή του κόστους το οποίο επομίστηκαν οι δημόσιοι φορείς που τις υποστήριξαν. Ο στόχος είναι ακριβώς να αντιμετωπίσουμε τη λεγόμε, τους λεγόμενους ηθικούς κίνδυνους, ώστε οι υπεύθυνοι που είναι για, τις, ε, για τους χρηματοπιστωτικούς αυτούς φορείς να μην επανέλθουν στις παλιές τους συνήθειες, στα σφάλματα του παρελθόντος, στην ε, αστοχία που υπήρξε σε ρυθμιστικό επίπεδο και το Κοινοβούλιο σας ήδη συζητά νέε ρυθμίσει για τα θέματα αυτά, είναι απαραίτητο να υπάρξει καλύτερο συντονισμό των εποπτικών και ρυθμιστικών δραστηριοτήτων, όπω γνωρίζετε πολύ καλά και εσεί ήδη. Χρειάζεται μια δράση από την πλευρά των υπευθύνων για την μακροοικονομική εποπτεία που δεν έλαβε χώρα πριν από την κρίση. Να γίνει καλύτερη αυτή λοιπόν η εποπτεία και μέσω των κανόνων εποπτείας από, τους, από τις ρυθμιστικές αρχές για τα χρηματοοικονομικά και μέσα από τις αρχές του ανταγωνισμού θα πρέπει να αποφύγουμε πρακτικές οι οποίες στο παρελθόν οδήγησαν στην κρίση που υφιστάμεθα σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δέχομαι την, ε, την ε, διόρθωση που κάνατε σε επίπεδο ονοματολογίας, αλλά είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που είναι σε πτώχευση ή όχι, νομίζω ήταν ανάλογη η κατάστασή τους χθες έλαβε χώρα μια συνάντηση όπου ήταν παρόν ο αρμόδιος για τη ρύθμιση στην Ιταλία, ο αρμόδιος της ε, Ιταλικής Τράπεζας, Κεντρικής Τράπεζας, κ. Καρουάνα, ο οποίος προειδοποίησε για ορισμένε πρακτικές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε υπερβολικούς κινδύνους για τις τράπεζες. Δεν σας ρωτώ περισσότερο για την τροποποίηση του πλαισίου εποπτείας, αλλά για το γεγονός ότι δόθηκαν κρατικές αρρωγές χωρίς καμία διάκριση και προς αυτούς οι οποίοι ήταν εσόφρονες και σε αυτούς που δεν ήταν εσόφρονες. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να τροποποιήσουμε το καθεστώς με το οποίο δίνονται αυτές οι αρρωγές προς το πιστοτικό ε, σύστημα, ώστε να πηγαίνουν μόνο στις ε, παρθένες οι οποίες είναι προσεκτικές και όχι σε αυτές οι οποίες ήταν μόρες ο κύριος Επίτροπος. Δεν γνωρίζω για το τελευταίο θέμα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι το πλαίσιο υποστήριξης για, το... για την αντιμετώπιση της κρίσης ήταν προσωρινό φυσικά και ένα προσωρινό πλαίσιο δεν μπορεί να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Τώρα πόσο μακρό διάστημα θα διατηρηθεί αυτή η μεταβατική κατάσταση, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα και μια πολύ δύσκολη και λεπτή απόφαση. Είναι πολύ εύκολο να πούμε σήμερα ότι μέσα σε χι μήνες έχει τελειώσει η κρίση. Αλλά τι θα γίνει μέσα σε αυτούς τους μήνες, μέσα σε έξι, μέσα σε οκτώ μήνες, τι θα γίνει στην πραγματική οικονομία. <clears throat> θα εκπληρωθούν οι πιο αισιόδοξε προβλέψεις ή θα επιβεβαιωθούν οι κασάνδρες. Εγώ πραγματικά δεν νομίζω ότι ξέρουμε. Έχουμε τόσο μεγάλο βαθμό αβεβαιότητος. Η κατάσταση μπορεί να είναι καλύτερη από ό,τι πέρσι αλλά εξακολουθούμε να κινούμεθα σε μεγάλη αβεβαιότητα και με μεγάλους κινδύνους για το χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Δεν θα ήταν υπεύθυνο από την πλευρά μου να πω ότι θα ακολουθήσουμε τον α ή β δρόμο. Όλα λοιπόν πρέπει να το πω ότι όλα είναι προσωρινά και όλα θα τελειώσουν κάποια στιγμή. Συγγνώμη που σας μπερδεύουμε με τα θέματα του χρόνου. Ξεχάσαμε να ανανεώσουμε το ορολόγιο και έτσι υπήρξε ένα πρόβλημα σε σχέση με τη χρονική αλληλουχία των παρεμβάσεων. Πάμε στον κύριο Μπάλτς τώρα. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αλμούνια και να τον καλωσορίσω. Έχω δύο ερωτήματα νομικά. Πρώτα απ' όλα για την εξέλιξη του δικαίου του ανταγωνισμού όσον αφορά την εξέλιξη του άρθρου 81 της ε, συνθήκης καθώς ξακολουθεί να μην έχει στο μέλλον δικαίωμα στην απόφαση στο Κοινοβούλιο. Μήπως ε, όμως ε, θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στη διαμόρφωση του δικαίου του ανταγωνισμού παρόλα αυτά. Δεύτερον, μιλήστε για την καταπολέμηση των καρτέλ, προβλεψιμότητα, διαφάνεια, όλα αυτά τα οποία ζητήσατε, αλλά νομίζω πως ε, όλα αυτά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα καθώς ε, δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση για αυτούς οι οποίοι θα είναι μάρτυρες εάν πρόκειται να καταθέσουν σε, κατά τέτοιων καρτέλ και δεν υπάρχει κάποια σύνθεση, σύνδεση μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών υπηρεσιών καταπολέμησης ε, των μονοπωλίων. Σκοπεύετε να κάνετε για αυτό το ζήτημα. Σε σχέση με το άρθρο 101, πρώην 81, γιατί πρέπει να μάθουμε τα νέα, τη νέα ρύθμιση των ε, άρθρων, Υπάρχουν διάφορες ε, διατάξεις, μιλάμε για εγκάρσιες συμφωνίες, δηλαδή ανακατηγορία, ως προς τις ε, συμφωνίες δηλαδή αυτές, όπου έγινε διαβούλευση με σας. Τώρα βεβαίως ε, εμβαθύνουμε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης, η ημερομηνία... μάλλον θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση πριν από το Μάιο. Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις του τομέα του, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των ασφαλιστικών εταιριών μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου. Έγινε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε σχέση με τις οριζόντιες συμφωνίες η προθεσμία για την αναθεώρηση είναι μέχρι τα τέλη του 2010. Θα τηρήσω αυτές τις ε, προθεσμίες και μπορώ να ακούσω και νέες γνωμοδοτήσεις ή να ανταλλάξουμε απόψεις μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι ότου λάβουμε αποφάσεις σε θέματα άκρο σημαντικά. Τόσο προς το δεύτερο ερώτημα για τους ε, υπεύθυνους εποπτείας για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τα καρτέλ, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε, διότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ακολουθήσουμε τους whistleblowers και από όσο γνωρίζω μέχρι τούδε, θα το δούμε βεβαίως αναπερίπτωση, αλλά από όσο γνωρίζω από την αρμόδια επίτροπο και από τη Γενική Διεύθυνση θα πρέπει να υπάρξει επίοικια τη στιγμή που υπάρχουν συγκεκριμένες ε, κατηγορίες και θα πρέπει έτσι να ορίσουμε την νέα πλαισίωση. Ε, ε, σύντομο ερώτημα για να επανέλθω. Μιλήσατε για τις ε, συλλογικές ε, προσφυγές. Με ποια βάση θα προωθεί κάτι γιατί βεβαίω είστε υπεύθυνο. Ε, θα είστε μάλλον υπεύθυνο για αυτό το, το ζήτημα νομίζω. Όπως σας, όπως σας είπα και πριν υπάρχουν διαφορετικές οδοί που μπορούμε να ακολουθήσουμε μέσα στα πλαίσια μιας συλλογικής αποζημίωσης. Διότι πολλές φορές η ζημία προκαλείται σε ΜΜΕ ή σε καταναλωτές διότι έγιναν καταχρήσεις από καρτέλ ή από δεσπόζουσα θέση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα και η αναγκαιότητα, θα έλεγα, να συμπληρώσουμε αυτή την αγωγή ως προς τις ε, ρυθμίσεις που υπάρχουν στον τομέα του ανταγωνισμού με αντίστοιχα μέτρα κύρωσης εξαιτίας της ζημίας που προκλήθηκε. Και αυτό μπορεί να γίνει δια της ιδιωτικής οδού. Δηλαδή, οι ζημιοθέντες μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση με διαδικασίες ε, μέσα στα πλαίσια και των ε, class actions των συλλογικών αγωγών γιατί υπάρχουν ε, ζημίες ε, κατά των, κατά των πολιτών καταναλωτών και κατά ΜΜΕ σε ορισμένες περιστάσεις. Ευχαριστώ. Τώρα προχωρούμε ε, προς την κυρία Γκύρι από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε σε ένα χαρτοφυλάκιο στο οποίο είναι απολύτως απαραίτητη η ανεξαρτησία, οπότε το ερώτημά μου αφορά ένα ζήτημα το οποίο έχει ζητηθεί πολύ στην Ουγγαρία το 2006 μετά τις βουλευτικές εκλογές σε μια συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών ο σοσιαλιστής Πρωθυπουργό ε, είπε πως ε, πράγματι είχαν κάνει τα πάντα ό,τι μπορούσαν στην προεκλογική εκστρατεία και ο Υπουργό ε, Οικονομικών είπε πω μετά από τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού ο κύριο Αλμούνια και οι συνάδελφοί του μα έδωσαν την ευκαιρία να συμπληρώσουμε το πρόγραμμα σύγκληση μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξή. Έχετε λάβει τέτοιο τηλεφώνημα από την Βουδαπέστη. ως αποτέλεσμα πολιτικής πίεσης συνταχθήκατε με τους σοσιαλιστές για να δώσετε έξι μήνες στην ε, κυβέρνηση για να συμπληρώσει το πρόγραμμα σύγκλησης ή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και το όνομά σας διασύρθηκε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καταρχήν. Ο, η Επίτροπος Ανταγωνισμού ο, ο Επίτροπος Ανταγωνισμού έχει κάθε δικαίωμα να ανοίξει ένα πολιτικό κόμμα και να έχει τις δικές του απόψεις. Οι δικέ μου απόψει είναι διαφορετικέ ίσω από την προηγούμενη Επίτροπο Ανταγωνισμού και από τον επερχόμενο Επίτροπο για τα Οικονομικά Θέματα. Δεν νομίζω ότι αυτό όμω θα επηρεάσει το έργο μα ω Επιτρόπων. Υπάρχει η πολιτική τη Κομισιόν, η οποία είναι μια εφαρμογή των συνθήκων και δεν έχει καμιά σχέση με προσωπικές, απο... προσωπικές απόψεις. Για την περίπτωση του 2006, από τη στιγμή που εγώ ήμουνα αρμόδιος για τα θέματα της, ε, τα οικονομικά και νομισματικά. Λίγες μέρες μετά από την ανάληψη καθηκόντων μου έγινε η διεύνηση και είχα πολλές συζητήσεις, πολλές επαφές για, με τους αρμοδίους γιατί δυστυχώς το δημόσιο έλλειμμα της Ουγγαρίας ήταν, πολύ, ήταν πάνω από το περίφημο 3% και χρειάστηκε το θέμα να παραπενθεί στο ΕΚΟΦΗΝ και να συζητηθεί και να υπάρξουν κάποιες προτάσεις προσαρμογής προς τις Ουγγρικές αρχές. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι πάντα στην Ουγγαρία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία σε οποιαδήποτε χώρα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν θέματα πειθαρχίας δημοσιονομικής, σε όλες τις περιπτώσεις εγώ εφάρμοσα τις συνθήκες, το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και επομένως μπορώ να σας πω ότι τώρα, επιτέλους, τα τελευταία χρόνια, οι ουγγρικές αρχές και η ουγγρική κοινωνία έχουν καταβάλει μια εξαιρετικά σημαντική προσπάθεια και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένο στο τέλος της θητείας μου Οικονομικού Επιτρόπου για το γεγονός ότι η Ουγγαρία <clears throat> έχει τηρήσει το πρόγραμμα το οποίο συνεφωνήθη και αυτό θα είναι μια βάση για την οικονομική ευμάρεια της Ουγγαρίας στο μέλλον να είναι επομένως τα πράγματα πολύ καλύτερα στην Ουγγαρία από ότι εάν δεν είχαν ακολουθήσει τις ε, συστάσεις που κάναμε βάσει του, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την απάντησή σας. Εγώ συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει και πολιτική ανεξαρτησία. Όλοι έχουν το δικαίωμα να έχουν την πολιτική οικογένεια στην οποία συμμετέχουν. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι για μας τους Ούγγρους είναι σαφές ότι η σοσιαλιστική κυβέρνηση παρουσίασε ψευδή στοιχεία και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δημοσιεύσουν τα στοιχεία που είχαν να κάνουν με το πρόγραμμα προσαρμογής, γιατί αυτά θα είχαν αποτέλεσμα στις εκλογές. Είπαν οι σοσιαλιστές ότι είχαν 2,4% έλλειμμα, ενώ ήταν 9%. Και έτσι κερδίσαν τις εκλογές. Και τις τελευταίες εβδομάδες στην ε, Ουγγαρία έλαβε χώρα μια απόφαση ενός δικαστηρίου που είπε ότι αυτή η απόκρυψη στοιχείων από την πλευρά της σοσιαλιστικής κυβέρνησης ήταν ε, αξιόπινη. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίσω ποια είναι η άποψή σας για αυτή την παράταση έξι μηνών για να παρουσιαστούν τα στοιχεία γιατί δόθηκε αυτή η παράταση έξι μηνών και μετά τις εκλογές επομένως. Ακολουθώ το... <laughs> την σύστασή σας, δεν θα εμπλακώ στην Ουγγρική πολιτική. Αλλά όταν μια χώρα έχει μια εκλογική διαδικασία είναι σαφές ότι οι δεσμεύσεις για την παροχή πληροφοριών για το πρόγραμμα προσαρμογής εκτός αν είναι νομικά απαιτητέ σε μία χρονική ημερομηνία όπως είναι τα στοιχεία για το έλμα όλα αυτά μπορούν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν στις εκλογικές αυτές αναγκαιότητες όταν προετοιμάζεται η ανάλυση εξουσίας από μια νέα κυβέρνηση. Νομίζω ότι στα πέντε χρόνια και κάτι που ήμουνα αρμόδιος ως Επίτροπος Οικονομικών Θεμάτων, μπορώ να σας δώσω ένα κατάλογο των περιπτώσεων όπου μια χώρα δεν έδωσε στη σωστή προβλεπόμενη ημερομηνία τα στοιχεία για την σύγκληση ή τη σταθερότητα λόγω εκλογικής διαδικασίας. Είναι μακροσκελέστατος αυτός ο κατάλογος, σας διαβεβαιώ. Ευχαριστούμε. Και τελευταία ερώτηση από το ΕΛΚ, ο κύριος Φεκμάρκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτός μικροφώνου κύριο κύριος Να το, το βρήκα το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ το ότι στις γραπτές σας απαντήσει τονίζετε πως είστε διατεθειμένος να λάβετε δράση κατά οποιασδήποτε εταιρεία κυβέρνησης παραβιάζει τους ζώο του ανταγωνισμού η προκάτοχός σας, η κυρία Νέλη Κρούς, επέβαλε ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα στην ιστορία, στην ε, τηλεφώνικα για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τι θα κάνατε εσείς σε αυτή την περίπτωση και πώς θα είχατε αντιδράσει και στις πιέσεις που θα είχατε οπωσδήποτε δεχτεί από την, ε, κυβέρνηση, από την κυβέρνησή σας. Κοιτάξτε, γνωρίζει η Ισπανική κυβέρνηση τι πίεση μπορεί να ασκήσει στον ε, Αλμούνια. Το ξέρουν πολύ καλά, μπορείτε να του ρωτήσετε. Ε, όσον αφορά την τηλεφώνικα, γεγονός είναι πως υιοθέτησε ένα πρόστιμο η Κομισιόν, αρκετά μεγάλο. Δεν θυμάμαι τώρα εάν η τηλεφώνικα ε, πήγε στο ΔΕΚ. Δεν θυμάμαι. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι πως πρέπει να παρακολουθήσουμε εάν ε, η στρέβλωση του ανταγωνισμού που ήταν αιτία του προστήμου εξακολουθεί να υφίσταται ή όχι. Και εξακολουθούμε να παρακολουθούμε τις εταιρείες και ειδικά τις μεγάλες εδρεωμένες εταιρείε που ήταν κρατικά μονοπόλια για το εάν συμμορφώνονται με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Αλλά να ε, επαναλάβω, τι θα είχατε κάνει εσείς. Θεωρείτε ότι ήταν σωστό αυτό το οποίο έκανε η προκάτοχός σας. Να επιβάλλει δηλαδή αυτό το πρόστιμο. Ε, είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση. Γιατί δεν ήμουν εγώ παρόν τότε. Είμαι μέλος του Σώματος των Επιτρόπων και ως μέλος της Επιτροπής υποστήριξα την απόφαση ανεπιφύλακτα. Ευχαριστώ. Προχωρούμε τώρα στους σοσιαλιστές και δημοκρατές. Την κυρία Αρλίν Μακάρθη. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είναι γεγονός ότι οι τράπεζες διεσώθηκαν από τα λεφτά των φορολογωμένων 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια παραπάνω από το ΑΕΠ της Γερμανίας και οι πολίτες έχουν εξοργιστεί ότι δόθηκε στις τράπεζες αυτές ένα τόσο μεγάλο ποσό και αυτό ουσιαστικά μείωσε και τον ανταγωνισμό λόγω τη κρίση. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω ποιε θα είναι οι δράσει που θα αναλάβετε ω Επίτροπο Ανταγωνισμού για να εξασφαλίσετε ότι ποτέ πια στο μέλλον ο, ο καταναλωτή, ο φορολογούμενος δεν θα πληρώσει την ύφη για την παράτολμη δράση των τραπεζών και θα ήθελα να με διαβεβαιώσετε ότι θα, ότι θα υποστηρίξετε οποιαδήποτε προτάση, έρθει στο Σώμα των Επιτρόπων για φόρο στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές ή για μια εισφορά των τραπεζών για να πληρώσουν οι τράπεζες ένα μέρος των σπασμένων. Και επίσης νομίζω το γεγονός ότι οι τράπεζες πληρώνουν υπέρογκα μπόνους αυτό είναι μια αποτυχία της πολιτικής ανταγωνισμούς. Και θα ήθελα να με διαβεβαιώσω ότι δεν χρησιμοποιηθούν δημόσιες επιδοτήσεις για να πληρωθούν μπόνους στα, στα μέλη του προσωπικού των τραπεζών. Η Κομισιόν, λέει ο κ. Επίτροπος, η Επίτροπη Μπαρόσο στην αρχή της ε, εντολής της, ενέκρινε μια σύσταση <clears throat> σε σχέση με τα συστήματα αμοιβών των υψηλών στελεχών. Μερικά χρόνια αργότερα, όταν ξεκίνησε η κρίση, αν θυμάμαι καλά, μόνο ένα κράτος μέλος ακολούθησε αυτές τις συστάσεις. Αλλά στην αρχή της κρίσης, λόγω του οικονομικού, της, της φάσης στον οικονομικό κύκλο και του υψηλού επίπεδου κινδύνου που βρεθήκαν σε αυτό πολλές ε, τράπεζες και πιστοτικά ιδρύματα λόγω των συστημάτων παροχής αμοιβών στα στελέχη τους, αυτό το θέμα δεν ήταν μονάχα στις ταπεινές προτάσεις της Κομισιόν, αλλά και στις προτάσεις του Οικονομικού Συμβούλιου και μέσα στις προτάσεις εποπτείας που έχουν αναφερθεί και ακόμα και σε επίπεδο G20 υπήρξαν σαφές, σαφείς λήψεις θέσεων για τα θέματα αυτά. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ευθύνε του Επιτρόπου Ανταγωνισμού, πράγματι όταν συζητούμε και αναλαμβάνουμε αποφάσεις για σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών που έχουν πάρει κρατικές επιδοτήσεις, εμείς θα εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά πώς χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα δημόσια κονδύλια που δόθηκαν ως επιδοτής και δεν θα δεχτούμε με τα δημόσια αυτά χρήματα που δόθηκαν για τη διάσωση αυτών των τραπεζών <clears throat> ή που υποστηρίχθηκαν αυτές οι τράπεζες θα μπορέσουν να πληρωθούν υψηλά μπόνους στα διευθύνοντα στελέχη τους. Και για το άλλο ερώτημα που θέσατε, ο φόρος στις οικονομικές συναλλαγές ή τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Εγώ έχω κάνει τους τελευταίους μήνες δημόσιες δηλώσεις, τονίζω ότι αυτό είναι μια καλή ιδέα. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσει κανείς αυτή την ιδέα, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα η οποία αξίζει την πλήρη προσοχή και συζήτηση μεταξύ όλων ημών. Σας ευχαριστώ. Μια περαιτέρω ερώτηση για τα χρηματοοικονομικά θέματα θα αναλάβετε να διερευνήσετε όπως κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις ΗΠΑ για να ξακριβώσετε αν υπάρχουν καρτέλ που λειτουργούν σε κέριους χρηματοοικονομικούς τομείς όπως παραδείγματος χάρη η αγορά, η αγορά ανταλλαγών ε, τα default swaps και άλλα τέτοια προϊόντα, χρηματοοικονομικά προϊόντα που δημιουργούν προβλήματα. Έχω δει αυτές τις πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς στην Ευρώπη, από την πλευρά της Κομισιόν, δεν έχουμε πάρει κανένα παράπονο <clears throat> προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά εξακολουθούμε να παρακολουθούμε και να αναλύουμε πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στις χρηματοοικονομικές αγορές σε αυτές τις δραστηριότητες που είναι εξόχως τεχνικές και πολυδέδαλες, αλλά που είναι πια πολύ πιο σημαντικές διότι έχουμε μάθει πολλά διδάγματα από την οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση. Αν υπάρξουν λοιπόν παράπονα προς την κατεύθυνση αυτή, σίγουρα θα τα εξετάσουμε τα θέματα αυτά. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμία τέτοια καταγγελία προς εμάς. Um, uh, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πιτέλα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Αν με συγχωρείτε, δεν σας είδα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αναγνωρίζουμε όλοι τις αρμοδιότητές σας ε, και τις δυνατότητές σας, ε, όπως διαπιστώνουμε και στη σημερινή ακρόαση. Εσείς είστε υπεύθυνο και για τον τραπεζικό τομέα. Θα ήθελα να σας μιλήσω και για τις τράπεζες λιανικής, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω έτσι, που ε, είναι επιζήμιες για τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές. Πώς μπορείτε να αποφύγετε κάτι τέτοιο. Siempre que a través με τα μέσα που διαθέτουμε ή από καταγγελίες όταν βλέπουμε ότι πρέπει να δράσουμε, αναλαμβάνουμε δράση. Αλλά σε αυτό τον ε, τομέα, πέρα από τις ε, δραστηριότητες ε, που ήδη γνωρίζετε. Δεν ξέρω κατά πόσο εσείς αναφέρεστε σε ένα άλλο νέο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Διότι ήδη με συναπόφαση έχουν ληφθεί ορισμένες αποφάσεις, αλλά βεβαίως ε, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα. Μιλώ ε, για διαφορετικές εισφορές. Υπάρχει και ένας κώδικας συμπεριφοράς για τις τράπεζες, και δεν ξέρω πώς θα επέμβεται. Συμφωνώ ως προς τον ανταγωνισμό, αλλά ο ανταγωνισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από κυρώσεις. Ως προς τις ε, κυρώσεις πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικέ, δηλαδή πέρα από τις ε, χρηματικές ε, κυρώσεις. Και για παράδειγμα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, κυρώσεις κατά διοικητών τραπεζών απάντηση στο σύστημά μας. Το σύστημά μας είναι ένα γερό, ε, στεναρό σύστημα, όπως είδαμε σε πολλές περιστάσεις. Και αυτό που έχει σημασία είναι να μην υπάρχουν υπεύθυνοι παρακόλλησης του ανταγωνισμού να δούμε πώς θα κινηθούμε στα πλαίσια των antitrust και ως προς τα κράτη θα πρέπει να δούμε πώς δρά το κάθε κράτος. Υπάρχει το θέμα των συλλογικών αποζημιώσεων που συζητούμε τώρα ως προς τις ε, κυρώσεις για πρακτικές κατά του ανταγωνισμού. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να μιλάμε μόνο για χρηματικές πίνες, αλλά και για άλλες ε, πίνε. Αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο φάσμα ενδεχόμενων αποφάσεών μας. Στον τομέα του ανταγωνισμού σε ορισμένες χώρες υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτω, στην πλειονότητα των χωρών που υπάρχει αυτή η δυνατότητα, 9 ε, χώρες από τις 27, είναι θεωρητική αυτή η δυνατότητα και μόνο σε μία χώρα έχει τεθεί στην πράξη. Άρα δεν μπορούμε να το συζητήσουμε τώρα, όμως δεν εντάσσεται στα πρότυπά μας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προβάλλουμε μια, ένα πρότυπο το οποίο έχει σταθεί αποδοτικό. Ε, πολλές φορές ε, βλέπετε ότι θέλω να σας σταματήσω. Ε, επόμενος, ο κύριος Σιμών, εξ Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Κύριε Επίτροπε, είχατε <clears throat> αναφερθεί στο θέμα της, των μεταφορών όπου υπάρχει ήδη πια μια ρύθμιση, η δυνατότητα ρύθμιση ε, από τη συνδίκη Λισαβόνα για τι κοινοφελεί υπηρεσίε. Η Επιτροπή Μπαρόσο είχε θέσει σαν κατευθυντήριε γραμμέ τη την εξασφάλιση ενό πλαισίου ποιότητα για τι ε, κοινοφελεί υπηρεσίε. Ο στόχο σήμαινε να είναι καλέ, προσιτέ και προσβάσιμε υπηρεσίε. Εγώ θέλω να θέσω τώρα δύο ερωτήματα σε σχέση με το θέμα αυτό και σα ευχαριστώ για την απάντησή σα. Πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο για την εξασφάλιση της σε ό,τι αφορά τι κοινωνικέ και κοινοφελεί επιχειρήσεις. Κατά την άποψή σα, ποιε θα μπορούσαν να είναι και οι, χρονικές, οι χρονικοί ορίζοντες για την εφαρμογή ενός τέτοιου πλαισίου ποιότητας. Χωρίς αμφιβολία συμφωνώ <clears throat> με αυτό το είπα το οποίο λέτε, όπως και προηγουμένως τόνισε ότι υπάρχει μεγάλη σημασία σε αυτό το τομέα. Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εργαστεί για το θέμα αυτό, η Κομισιόν έχει σκεφτεί ιδιαίτερα για το θέμα αυτό και υπάρχουν στις συνθήκες νέες <clears throat> ρήτρες και μια νέα νομική βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε και να οδηγήσουμε σε στο να κατασταλάξει η ανάλυση προς το πρακτικό επίπεδο. Τώρα, πώς βλέπω τη διαδικασία λήψης απόφασης. Καταρχήν, όπως ξέρετε, και ελπίζω θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και στους επόμενους μήνες, προετοιμάζουμε μια αξιολόγηση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι δημόσιες επιδοτήσεις σε σχέση με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Αυτό υπήρχε ήδη σαν δέσμευση από την πλευρά της Κομισιόν. Υπάρχει η αλλαγή ...τη συνθήκης, το νέο κοινοβούλιο, η νέα επιτροπή και γι' αυτό προτιμούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τα θέματα αυτά το, μέσα στο 2010 και <clears throat> όχι αυτή τη στιγμή να το κάνουμε προηγουμένως. Βέβαια, υπάρχουν πολλές οπτικές γωνίες, δεν είναι μοναχά θέμα ανταγωνισμού υπάρχουν και άλλες πτυχές, άλλες πολιτικές ευρωπαϊκές όπου θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την η στοχοδεσία τους για τις υπηρεσίες κοινοφιλούς ενδιαφέροντος να υλοποιηθούν στην πράξη. Και τέλος υπάρχει μια μεγάλη πολυμορφία σε, στις υπηρεσίες αυτές και στις χώρες μας. Υπάρχει διαφορετική σύλληψη του τι είναι μια κοινοφελής υπηρεσία ή του τι είναι μια μη οικονομικού χαρακτήρα κοινοφελής ε, υπηρεσία. Δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο αυτή η διάκριση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και το νομικό θέμα και εσείς αναφέρατε το άρθρο 14 και το άρθρο 106 των συνθηκών αναφέρεται στην, ε, στις κοινοφελείς υπηρεσίες και είναι νομική βάση για τη δράση της Κομισιόν στα θέματα αυτά. <clears throat> Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πιανού ίδιους ρυθμιστικό πλαίσιο είναι απαραίτητο και αυτό ακριβώ ήθελε να επιτύχει ο πρόεδρος Μπαρόσο στι κατευθυντικέ γραμμές και να υπάρξει μια ευρεία συνένεση γιατί τα θέματα αυτά είναι σημαντικά και για το υπόδειγμα κοινωνίας μας. Δεν είναι μόνο μια οικονομική συζήτηση, είναι θέμα κοινωνίας επίσης. Ευχαριστώ. Τα τελευταία χρόνια θέλω να σας πενθυμίσω το θέμα αυτό επηρεάστηκε και από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και είναι απαραίτητο εδώ πέρα να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτή η Κομισιόν, πώς, να, πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πολυμορφία την οποία αναφέρατε κι εσείς, πώς θα αποφύγουμε να φτάσουμε σε μια ρύθμιση η οποία θα είναι μονάχα ο κατώτερος κοινός παρανομαστής σε επίπεδο ποιότητας. Συμφωνώ, υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ένα τέτοιο πλαίσιο. Το είπε και ο πρόεδρο Μπαρόσο, το είπα και εγώ και πολλοί από του συναδέλφου μου σε αυτέ τι ακροάσει οι οποίε γίνονται αυτή τη βδομάδα. Το πραγματικό ερώτημα είναι. Χρειάζεται για να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο να κατέλθουμε στο χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Μέχρι ποιου βαθμού είναι αυτό πρόσφορο να έχουμε απλώς ένα ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Υπάρχουν πολλές φορές ρυθμίσεις τομεακές. Σε ορισμένους τομείς υπάρχει ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε άλλες περιοχές δεν υπάρχει τέτοια ρύθμιση. Δεν είναι εύκολο το ερώτημα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από πολιτική έποψη. Είναι λεπτό και δύσκολο, αλλά πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Σίγουρα δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Μεταξύ της επιζήτησης μιας οριζόντιας ρύθμισης και της φιλοδοξίας να υπάρχει ρύθμιση σε υψηλό επίπεδο θα πρέπει να καταλήξουμε να βρούμε κάποια ισορροπία. Ε, Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα σε κάποιες ερωτήσεις από τους φιλελεύθερους. Πρώτα απ' όλα η Σόφη Ινετφέλτ. Ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλωσορίζω την διάθεση συνεργασίας που δείχνετε με το Κοινοβούλιο. Αναμένω αυτή τη συνεργασία, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να αντιμετωπίσετε και τα κράτη-μέλη, που μπορεί να μην είναι τόσο συνεργάσιμα όσο το Κοινοβούλιο. Και σε καιρούς κρίσης ε, φύσανται πίεση οι πολιτικές του ανταγωνισμού, ειδικά από τα προστατευτικά αντανακλαστικά των κρατών μελών που θέλουν να δώσουν κρατικές ενισχύσεις και κάποιες κυβερνήσεις και κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα τείνουν να παρουσιάζουν τους κανόνες του ανταγωνισμού ως ε, ζουρλομανδία για τις εθνικές ε, πολιτικές, ως στενό κορσέ μάλλον καλύτερα. Πώς θα ξεπεράσετε την απροθυμία να περιοριστούν αυτά τα σχέδια κρατικών ενισχύσεων, πώς θα οδηγηθείτε σε ανάκτηση παρανόμων κρατικών ενισχύσεων, στις οποίες κάποια κράτη-μέλη είναι υπότροποι. Και ανέφερε και η κυρία Γκουλάρ κάτι παρόμοιο, πώς θα πείσετε τα κράτη-μέλη να σταματήσουν να κατηγορούν συνεχώς τις Βρυξέλλες και να ξεκαθαρίσουν στην κοινή γνώμη πως η επιβολή των κανόνων του ανταγωνισμού είναι σημαντική για την προστασία των καταναλωτών και την υγεία της οικονομίας. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω πως το τμήμα της απάντησης στην ερώτησή σας θα είναι η έκθεσή σας. Ε, δηλαδή πρέπει να μας βοηθήσει. Να βρούμε τα σωστά επιχειρήματα για να εξηγήσουμε στους πολίτες μας γιατί χρειάζεται ο ανταγωνισμός για να διατηρήσουμε την εσωτερική αγορά, για να δημιουργηθούν οι συνθήκες ε, βιώσιμης ανάπτυξης, ε, ανταγωνιστικής οικονομίας, για στιβαρές εταιρείε κτλ. κτλ. Τώρα, για την κοινή γνώμη στο ζήτημα αυτό, αφενός η Κομισιόν είναι κατά κύριο υπεύθυνη για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, οπότε πρέπει να είναι αυστηρή και δίκαια, να υπάρχει ίση μεταχείριση, οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται την Κομισιόν ως αμερόληπτη και αυστηρή, και ταυτόχρονα πρέπει να εξηγούμε. Πρέπει να πείσουμε. Να δίνουμε καλά παραδείγματα. Και έχουμε φανταστικά παραδείγματα στην Ευρώπη για το πώς η απελευθέρωση και ο ανταγωνισμός δημιουργεί ωφέλη για τους πολίτες. Αν δούμε τώρα τις φρινές πτήσεις, ε, τις τηλεπικοινωνίες, μπορούμε να εξηγήσουμε πολλά πράγματα. Και όταν συζητάμε τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού στο εθνικό επίπεδο, τα προβλήματα με τις ε, τιμές των τροφίμων σε κάποιους τομείς. Έχουμε λαμπρά παραδείγματα. Οπότε, δίκαιοι, αμερόληπτοι και ταυτόχρονα και πολιτικά επιχειρήματα και επικοινωνία και διάλογος με τους πολίτες. Νομίζω αυτή είναι η συνταγή. Όσον αφορά τώρα την ανάκαμψη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, το ποσοστό κρατικών ε, ενισχύσεων, των ασύμβατων κρατικών ενισχύσεων που έχει ανακτηθεί, αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. Στις αρχές της δεκαετίας που μας πέρασε ήταν γύρω στο 25% των συνολικών ασύμβατων κρατικών ενισχύσεων, όπως τις έκρινε το Δικαστήριο και η Κομισιόν, και τώρα είναι 90%. Ε, Ξέρω πως εκκρεμούν ακόμα γύρω στις 50 ε, υποθέσεις, αλλά σκοπεύω να αυξήσω το 90%. Θέλετε να επανέλθετε γρήγορα, Σόφη. Όχι, εντάξει. Ωραία, περνάμε στον Καρλ Χάγκλουντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, να ρωτήσω την άποψή σας για την πολιτική του 2020. Βασική σας πολιτική είναι να δημιουργηθεί μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη και ως υπεύθυνο για την πολιτική ανταγωνισμού. Πώς θεωρείτε πως μπορεί να συνεισφέρει πολιτική ανταγωνισμού στην, πολιτική, στην επιτυχία αυτής της πολιτικής και επιπλέον ε, πώς θα λέγατε ότι μπορεί να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης έναντι των ΙΠΑ ε, στο διεθνές επίπεδο. Η στρατηγική 2020 ε, είναι ακόμα ένα ερωτηματικό. Προετοιμάζουμε την συζήτηση, το Συμβούλιο της 11 Φεβρουαρίου θα το συζητήσει αυτό στο επίπεδο των αρχηγών κρατών με τον πρόεδρο της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν ξέρω επί τη ευκαιρία αν ε, είναι προσκεκλημένος ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Μετά από αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η νέα Επιτροπή Καλό χόντων των πραγμάτων, θα προετοιμάσει μια πρόταση για το Εαρινό Συμβουλίο του Μαρτίου. Ποιος είναι ο ρόλος ε, της ε, στρατηγικής ε, ανταγωνισμού για να έχουμε πιο ανταγωνιστική, πιο βιώσιμη οικονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικός γιατί αν δεν λειτουργούν επαρκώς οι αγορές μας δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί ούτε στην εσωτερική αγορά ούτε ως προς τους εταίρους μας στην παγκόσμια οικονομία και χωρίς επαρκή χρήση δημοσίων κονδυλίων για να ενθαρρυθούν κάποιες δραστηριότητες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πράσινες δραστηριότητες, ε, εκπαίδευση, κατάρτιση, δεν θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως όλες τις ε, δυνατότητες ε, που θα έχουν οι κυβερνήσει. Αυτά είναι δύο στοιχεία κλειδιά για τη στρατηγική του 2020, όχι τα μόνο αυτά, αλλά και επίσης γίνεται μια συζήτηση τουλάχιστον στη χώρα μου αυτή τη στιγμή και σε άλλες χώρες. Διάβασα στον τύπο πως θα πρέπει η στρατηγική αυτή να είναι δεσμευτική, λιγότερο δεσμευτική. Κοιτάξτε, η πολιτική του ανταγωνισμού έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, είναι δεσμευτική. Να επανέλθω λίγο σύντομα ε, μετά την καλή απάντηση του κ. Πιτρόπου μετά τη συζήτηση που μόλις είχαμε για τις κρατικές ενισχύσεις και την κρίση. Θεωρείτε πως ε, θα πρέπει να οδηγηθούμε σε κάποιο πιο έτσι, συνεκτικό πλαίσιο αντιμετώπισης μελλοντικών κρίσεων και πώς θα το ενσωματώσετε αυτό στην πολιτική ανταγωνισμού και σε τυχόν ε, μελλοντική στρατηγική. Βλέπετε να υπάρχει κάποια σύνδεση. Δεν υπάρχει Η σύνδεση. Η διαχείριση των κρίσεων, ιδίω στην εσωτερική μας αγορά, όταν έχουμε 40 ή 45 διαμεθοριακές, διαμεθοριακά τραπεζοπιστωτικά ιδρύματα που είναι καρδιά του συστήματος μας, προφανώς είναι κεφαλαιώδης η διαμεθοριακή διαχείριση των κρίσεων. Χωρίς αυτή θα επαναλάβουμε απλώς τα προβλήματα που έχουμε περάσει τα δύο προηγούμενα χρόνια για να λύσουμε τα προβλήματα μονάχα ορισμένων φορέων και κανόνε άλλου. Ο σύνδεσμο τώρα με την πολιτική ανταγωνισμού δεν είναι άμεσο. Αν η διαχείριση τη κρίσεω είναι αποτελεσματική και επαρκή, υπάρχει λιγότερη δουλειά σε ό,τι αφορά την ε, διάσωση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και λιγότερες κρατικές επιδοτήσεις, αλλά δεν βλέπω καμία άμεση σύνδεση βλέπω μια σύνδεση μεταξύ της διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και του επίπεδου ε, πόρων που δίνονται στα ευρωπαϊκά χέρια. Γιατί χωρίς ευρωπαϊκούς πόρους είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό που έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές στο ΕΚΟΦΗΝ για την κατανομή του άχθους. Αν πρέπει λοιπόν να διασώσετε ή να βοηθήσετε διαμεθοριακά ιδρύματα και η χρηματοδότηση είναι μόνο εθνική θα έχουμε πολύ δύσκολες συζητήσεις. Προχωρούμε τώρα στους πράσινους και στον κύριο Κέντεν. Ευχαριστώ κύριε Αλμούνια. <clears throat> Καλησπέρα καλύτερα. Υπήρξατε επίτροπος στην Επιτροπή του 2004 πριν από την κρίση και αναγκαστήκατε να πάρετε κάποιες αποφάσεις οικονομικού χαρακτήρα. Σήμερα ουσιαστικά ανανεώνουμε την εμπιστοσύνη που σας δίνουμε ως νέο επίτροπο με νέο χαρτοφυλάκιο. Η κρίση οικονομική, η χρηματοοικονομική αυτή άλλαξε τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. Ποιες αποφάσεις πήρατε μεταξύ του 2004 και του 2008 που τώρα μετανοείτε για αυτές τι είναι αυτό το οποίο δεν θα κάνατε πια, υπάρχει κάτι για το οποίο μετανοείτε, υπάρχει κάποιο στοιχείο του απολογισμού που μπορείτε να κάνετε για το παρελθόν, για το οποίο θέλετε να γίνει κάποια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο δράει η Κομισιόν. Ως πολιτικός δεν <clears throat> μιλώ, δεν είμαι συνηθισμένος να μιλώ δημόσια για τις αποτυχίες μου περισσότερο προτιμώ να μιλάω για τις επιτυχίες μου. Πιστεύω, μεταξύ άλλων, μεταξύ άλλων επιτυχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν, σε σχέση με την αντιμετώπιση των κρίσεων, υπήρξε ένα πολύ καλό παράδειγμα καλή αντίδραση προ την κρίση από την Κομισιόν, από την Κεντρική Τράπεζα, από τις κυβερνήσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά όμως, νομίζω ότι η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητα και ανάπτυξη το 2005, όπου εγώ πήρα την πρωτοβουλία το Σεπτέμβριο 2004 να αποκαλέσω αυτήν την ε, ε, συζήτηση μέσα στους τελευταίους μήνες της Επιτροπής πρώτη, αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό για να μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας, το οποίο να είναι αρκετά ευέλικτο σε στιγμές βαθιάς κρίσης όπως αυτή που γνωρίσαμε τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτά είναι τα θετικά. Για τα λιγότερα θετικά τώρα, νομίζω ότι είναι προφανές ότι η στρατηγική της Λισαβόνας, την οποία αναθεωρήσαμε το 2005, δεν κινήθηκε επαρκώς προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν είχε αρκετά ισχυρά εργαλεία για την παρακολούθηση και την εφαρμογή των στόχων της στις κύριες πολιτικές αυτής της στρατηγικές. Το 2005 ήταν ένα έτος όπου η ευρωπαϊκή οικονομία παρεχόταν μετά από μια ύφεση 2002-2003 στην οικονομική ανάπτυξη. Είχαμε την ε, ε, εμπειρία του διαστήματος 2000 με 2005 για την έλλειψη αποτελεσμάτων από την αρχική <clears throat> στρατηγική της Λισαβόνας. Συζητήσαμε, επιφορτήσαμε το Βιμ Κοκ και μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με το να συντάξουν μια έκθεση που ήταν πολύ καλή, αλλά δεν καταφέραμε το Μάρτιο 2005 να πείσουμε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να δώσουν πιο δεσμευτικά εργαλεία εφαρμογής στρατηγικής Λισαβόνας. Και νομίζω τώρα πια δεν πρέπει να επαναλάβουμε αυτό το σφάλμα. Μεταξύ των κρίσεων που γνωρίζουμε υπάρχει μια κρίση του περιβάλλοντος, η κρίση της κλιματικής αλλαγής. Εγώ θα ήθελα να ξέρω εσείς ως επίτροπος που είσαστε υπεύθυνος για την πολιτική ανταγωνισμού πώς θα ενσωματώσετε τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, <clears throat> της σχέσης ενέργειας και κλίματος. Όλα αυτά έχουν κάποια σχέση με την πολιτική ανταγωνισμού ή η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να σέβεται και τα διακυβεύματα του περιβάλλοντος. Νομίζω ότι έχει βελτιωθεί το πλαίσιο ενσωμάτωσης. Όταν όμως δούμε την ε, τομιακή προσέγγιση, όπως έγινε από την Έλλη Κρούς, από την προκάτοχό μου, βλέπουμε ότι ένα μέρος έχει ενταχθεί στο πακέτο ενέργειας και ένα άλλο στις ε, νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ του περιβάλλοντος. Όλα αυτά μπορούν να βελτιωθούν, διότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ε, κλιματικές αλλαγές. Αυτό αποτελεί ε, βασική κατευθυντήρια γραμμή και γι' αυτό θα πρέπει να κινηθούμε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη από πλευράς περιβάλλοντος και άρα και η πολιτική ανταγωνισμού και από άποψη αντιτράστ και από άποψη κρατικών ενισχύσεων και ρύθμισης τους θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτή την πλαισίωση. Και στον τομέα της ενέργειας ή στις ε, περιβαλλοντικές κρατικές ενισχύσεις έχουμε συνεισφέρει και θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε όλο ένα και περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, από τον κύριο Γκίγκολτ είναι η επόμενη ερώτηση. Καλώς ήρθατε. Κύριε Ελμούνια, χαίρομαι που σας ε, ξαναβλέπω. Έχω ένα ερώτημα όσον αφορά τον φορολογικό ανταγωνισμό. Είστε αρμόδιος και για την ρύθμιση στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Πολλά κράτη-μέλη δίνουν έμεσα κρατικές ενισχύσεις μέσω κάποιων φορολογικών ευεργετημάτων και αυτό είναι πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό και αναρωτιέμαι αν είστε διατεθειμένος να χρησιμοποιήσετε τα μέσα που έχετε στην διάθεσή σας για να καταπολεμήσετε αυτή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού καθώς είναι μια πλάγια παρέμβαση στον ανταγωνισμό μέσω φορολογικών ε, ευνοημάτων, ευεργετημάτων. Όπως, όπως πριν απάντησα και στον κύριο Λαμπέρ, υπάρχουν περιορισμοί. Δεν μπορώ να κινηθώ πέραν των περιορισμών που ορίζουν οι συνθήκες. Οι συνθήκες ορίζουν ότι μπορούν να υπάρξουν φορολογικές ρυθμίσεις οι οποίες είναι συμβατές. Εάν λοιπόν μέσω φοροελαφρύνσεων δεν δίνουμε κίνητρα για την βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος ή εάν τασόμαστε υπέρ ε, μορφών ενέργειας που δεν είναι ανανεώσιμες, θα δράσουμε όπως πρέπει να δράσουμε, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Έχω την ε, εντύπωση ότι ε, δεν υπήρξε καλή κατανόηση του ζητήματος. Οι προκάτοχοι σας ε, χρησιμοποίησαν την νομοθεσία, την ομοθέσια κατά των κρατικών ενισχύσεων για να ρυθμίσουν θέματα ανταγωνισμού. Άρα εσείς έχετε στη διάθεσή σας αυτά τα μέσα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε κατά πόσο υπάρχει ρυθμιστικό ε, πλαίσιο ή διακριτική ευχέρεια και τι μπορείτε να κάνετε στα πλαίσια της συνθήκης έτσι ώστε να περιορίσετε τις τρευλώσεις του ανταγωνισμού και της αγοράς. Δηλαδή, νομοθεσία κατά των κρατικών ενισχύσεων, τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καταπολεμήσετε την στρέβλωση του ανταγωνισμού και ενισχύσεις που να βασίζονται στη φορολογία. Προς επιχειρήσεις, ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Σας είπα αρχικά ότι θα αναλάβω ε, μέτρα, θα δράσω στα πλαίσια της συνθήκης. Και το, το ίδιο είπατε και εσείς στη δευτερολογία σας, άρα συμφωνούμε απόλυτα. Τώρα ο κύριος Μπόκρος έχει το λόγο από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αλμούνια, υπό το παρόν χαρτοφυλάκιο, μάλλον ε, με βάση τα καθήκοντά σας μέχρι τώρα, είχατε την δυνατότητα να συνεργαστείτε με πολλούς φορείς, μερικοί και μερικές χώρες διανύουν μεγάλη κρίση. Ε, ορισμένες χώρες είναι πιο ανταγωνιστικές από αρκετές ε, δυτικές χώρες και μπορούν να ρυθμίσουν καλύτερα τους κανόνες ανταγωνισμού. Όταν λοιπόν ε, έγινε λόγος για έλλειψη συσχετισμού μεταξύ διαχείρισης κρίσεων και πολιτικής ανταγωνισμού, αναρωτιόμουν κατά πόσο έχουμε να μάθουμε πολλά από την πρακτική και από την πείρα αυτών των χωρών που δεν είχαν τα φορολογικά μέσα για να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό, μη έχοντας τη δυνατότητα ε, να εφαρμόσουν συγκεκριμένα προγράμματα. Ε, για παράδειγμα απόσυρσης. Δηλαδή είναι μερικοί, μερικές χώρες οι οποίες είναι καλύτερα ρυθμισμένες για να αντιμετωπίσουν θέματα ανταγωνισμού γιατί σε ορισμένες ε, ανατολικές ε, χώρες δεν έγινε λόγος για εθνικούς πρωταθλητές οι οποίοι ε, την χάνουν υποστήριξη σε μια περίοδο κρίσης. Ποια είναι τα διδάγματα που λάβαμε από αυτές τις χώρες και που θα ήταν ε, σκόπιμο να χρησιμοποιήσετε στο, στα νέα σας καθήκοντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έμαθα πολλά κατά τα πεντέμιση αυτά χρόνια ως προς τις οικονομικές προτεραιότητες και στάσεις, καθώς και τον ορισμό φορολογικών και άλλων ε, πολιτικών, όπως ε, από χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Έχουμε να κάνουμε με δύο περιόδους, πριν από την κρίση και κατά την κρίση. Πριν από την κρίση ήταν άκρος εντυπωσιακό διότι θυμάμαι ότι με τον όλη Ρεν που θα ασχοληθεί με οικονομικά και νομισματικά ζητήματα τώρα, μιλήσαμε για τα, πρώτα, για τα πρώτα πέντε χρόνια της διεύρυνσης και δώσαμε μια θετική ανάλυση με δυναμισμό που διέπεται από δυναμισμό, κίνητρα για μεταρρυθμίσεις και βελτίωση ΑΕΠ, κατακεφαλή ΑΕΠ, κράτους προνοίας, καθώς και ε, νέες επενδύσεις. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, τα χρόνια της ε, κρίσης, η αποτίμηση είναι κάπως διαφορετική. Αυτό που οφείλεται, οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάπτυξη αυτών των χώρων σε διαφορετικά επίπεδα αλλά υπάρχει ένα γενικό χαρακτηριστικό που διέπει τις ε, χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ένα μέρος της ανάπτυξης οφειλόταν στις επενδύσεις από το εξωτερικό που τώρα έχει εκλείψει. Επίσης είχαν πολλά έσοδα από εμβάσματα από μετανάστες και οι εξωτερικές αγορές για τις εξαγωγές τους δηλαδή μειώθηκαν Άρα οι αδυναμίες αυτού του αναπτυξιακού μοντέλου φάνηκαν, διαφάνηκαν και έφτασαν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ήθελα να πω ότι ο τρόπος διαχείρισης των κυβερνήσεων πριν από την κρίση ήταν πολύ σημαντικός για την αντιμετώπιση της μεταγενέστερης κρίσης. Είχαμε καλές αλλά και κακές περιπτώσεις σε αυτές τις χώρες. Χώρες που θα ανακάμψουν και που θα είναι πολύ δυναμικές εκ νέου κατά τα επόμενα χρόνια. Ε, πολύ σύντομη η δευτερολογία. Το ζήτημα είναι κατά πόσο υπάρχουν ε, επιπτώσεις ως προς το νέο σας ε, χαρτοφυλάκιο, αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή στο ως προς τη, τα καθήκοντά σας στο τομέα του ανταγωνισμού δεν μπορώ να διακρίνω τη μία χώρα από την άλλη ως Επίτροπος Επιθεμάτων Ανταγωνισμού. Υπάρχει νομοθεσία περί ανταγωνισμού, οι συνθήκες, οι διατάξεις των συνθήκων που ισχύουν σε όλες τις χώρες. Δεν μπορώ να προβώ σε διάκριση. Δεν μπορώ να ε, πω στους ανθρώπους από πού προέρχονται για να είμαι πιο ευέλικτος ή πιο αυστηρός, πιο επίκης ή πιο αυστηρός. Οι πλουσιότερες χώρες έχουν περισσότερες δυνατότητες να χρησιμοποιήσουν τις κρατικές ενισχύσεις. Οι μεγαλύτερες οικονομίες, οι πιο πλούσιες οικονομίες είχαν μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν το δέλεαρ να χρησιμοποιήσουν τη δεσπόζουσα θέση ή να την καταχραστούν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, το πλαίσιο θα πρέπει να ισχύει και στα 27 κράτη-μέλη. Ο κύριος Φόξ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αλμούνια, <clears throat> θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με τα πρόστιμα τα οποία εφαρμόζει η Κομισιόν για μη ανταγωνιστικές πρακτικές σε εταιρείε. Τι πρέπει να γίνεται με τα χρήματα τα οποία συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι πρέπει να επανέρχονται στα κράτη-μέλη και εάν ναι, με, εάν, εάν ναι, πώς θα τα κατανείμετε για να αποζημιώσετε μερικά κράτη-μέλη τα οποία επλήγησαν περισσότερο από αυτές τις αντιανταγωνιστικές ε, πρακτικές. Θα ακολουθήσετε μια κλίδα πληθυσμού, μια κλίδα συμμετοχής στον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και αν πιστεύετε ότι πρέπει να έρθουν στα κράτη-μέλη τα χρήματα αυτά, με ποιο τρόπο πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν υπάρχει η διαδικασία προσφυγής κατά των προστήμων, αλλά στη συνέχεια γίνονται πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε, όταν υπάρξει πλεόνασμα στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το πλεόνασμα επανέρχεται στα κράτη-μέλη βάσει της ίδιας κλίδας κατανομής που χρησιμοποιείται για τη συνεισφορά των κρατών μελών στον προπολογισμό. Αλλά οι πόροι αυτοί μπαίνουν στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πόροι από τα πρόστιμα. Σαν παράδειγμα, <clears throat> ας υποθέσουμε ότι μία πρακτική που παραβιάζει τον ανταγωνισμό αφορούσε ιδιαίτερα την Ισπανία. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα, με περισσότερη αποζημίωση προς την Ισπανία <clears throat> από την πρόσοδο αυτών των προστήμων. Θεωρείτε λοιπόν ότι το σύστημα που ισχύει τώρα είναι επαρκές για να αποζημιώσει τα κράτη-μέλη που θίγονται από αυτές τις πρακτικές. Είσαστε ικανοποιημένος με την τωρινή κατάσταση. Όχι. Είτε είναι η Ισπανία, είτε είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε είναι οι κάτω χώρες, οποιαδήποτε χώρα και να είναι, δεν μπορούν να ζητήσουν να πάρουν τα χρήματα για αυτούς. Τα χρήματα αυτά ανήκουν στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συζητήσουν μαζί με το Κοινοβούλιο πώς γίνονται οι δαπάνες του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές ελπίζω ότι θα ανταρακλώνται καλύτερα προτεραιότητες της Ευρώπης από τις τις Ο κ. Κλούτ για την Γκουε έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ο συνάδελφος κ. Σέντλ ήθελε να κάνει την ερώτηση, οπότε τον αντικαθιστώ εγώ γιατί αρρώστησε. Κύριε Αλμούνια, στις γραπτές σα απαντήσει. είπατε πω το Δεκέμβριο του 2008 θεωρήσατε πως θα πρέπει να εισαχθούν περαιτέρω μέτρα όσον αφορά τις ε, κρατικές ε, ενισχύσεις. Αυτό αφορά την ε, μεταφορά εργοστασίων όπως παραδείγματο χάρη από την Ιρλανδία στην ε, Πολωνία εντός της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με άλλα λόγια θα βρει επιτέλους ε, το θάρρος ε, η Κομισιόν να επιβάλλει ένα τέλος μεταφοράς τέτοιων εργοστασίων για να σταματήσει αυτή η διαδικασία. Εγώ προέρχομαι από το Ρούργκεμπιτ, μεγάλη βιομηχανική περιοχή και μπορώ να σας πω πως υπάρχει πράγματι αυτός ο ανταγωνισμός ε, όσον αφορά το που θα πάνε τα εργοστάσια, Opel, τα ξέρετε, μεταξύ δηλαδή του Bochum και λοιπόν σημείων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σε σχέση με το πρώτο τμήμα της ερώτησής σας, σε σχέση με το, τα χρονικά περιθώρια της ενίσχυσης μη χρηματοδοτικού τύπου που εισήχθη στο τέλος του 2008, πρόκειται για κάτι που θα ισχύσει μέχρι το τέλος του 2010 αυτή είναι η προθεσμία, αλλά αυτή, αυτή την προθεσμία θα πρέπει να την επιβεβαιώσουμε ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες. Πρόκειται για μια εξαίρεση για να αντιμετωπίσει την ε, κρίση, όχι για την πτώση της κυκλικής ε, τακτικής δραστηριότητας. Εάν βρισκόμαστε εκτός ε, κινδύνων, με βάση την κρίση που διανύουμε τώρα, θα τηρήσουμε την προθεσμία, δηλαδή μέχρι τα τέλη του 2010, όπως ίσχυε με τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά εσείς αναφερθήκατε στην ΤΕΛ. Μπορώ να σας πω χωρίς να είμαι ειδικό, ότι δεν υπάρχει μία ε, μηχανιστική σχέση αυτού που αποφώσει η Επιτροπή για την ΔΕΛ στην Ιρλανδία σε σχέση με την ΔΕΛ στην Πολωνία. Πρόκειται για δύο διαφορετικά επενδυτικά προγράμματα. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας χρησιμοποιήθηκε το Ταμείο ε, Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, χρησιμοποιήθηκε αυτό το κονδύλιο για την Ιρλανδία και στην περίπτωση της ΔΕΛ της ε, Πολωνίας ε, πρόκειτο για κρατική ενίσχυση ως προς μία επένδυση που δεν σχετίζεται με την επιχείρηση της Ιρλανδίας δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να μην άπτεται αυτή τη ενίσχυση ή που αυτή η ενίσχυση να μην είναι συμβατή με το πλαίσιο της ΔΕΛ. Αν μου επιτρέπετε να επανέλθω από πλευράς ε, εργαζομένου. Το ζήτημα είναι πως ε, πηγαίνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μεταφέρονται εργοστάσια και δεν ε, δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Εάν γίνονταν κάτι τέτοιο δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να μιλάμε για μεταφορά εργοστασίων απλά. Και ουσιαστικά μιλάμε για ανταγωνισμό μισθοδοσίας, αν θέλετε, μεταξύ Πολωνίας, Ιρλανδίας και τα λοιπά και εδώ είναι και το ζήτημα της φορολογίας. Πώς θα σταματήσει αυτός ο κοινωνικός ανταγωνισμός. Ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το δούμε επικριτικά, γιατί έτσι τελικά οι εργαζόμενοι καταλήγουν να είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως υφίσταται και αυτή η πίεση μέσω των πολιτικών επιδότησης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατανοώ απόλυτα τα επιχείρηματά σας. Σας λέω όμως ότι δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι δεν υπάρχει συσχετισμός, άμεσος συσχετισμός μεταξύ της, ε, του κλεισίματος ενός εργοστασίου μιας επιχείρησης και του ανοίγματο σε μία άλλη χώρα που μπορεί να λάβει αυτές τις ενισχύσεις γιατί τότε οι Πολωνοί θα έπρεπε να ρωτήσουν γιατί αυτή, η, αυτή την ενίσχυση που έχω δικαίωμα να λάβω δεν λαμβάνω σε αυτήν την περίπτωση. Ποιος είναι ο λόγος θα μας ρωτούσαν οι Πολωνοί. Δεν υπάρχει όμως συσχετισμός του κλεισίματος ενός εργοστασίου που μας σε ιδιαίτερα και εδώ θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους ε, εργαζόμενους μέσα στα πλαίσια του Ταμείου ε, Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης και της άλλης περίπτωσης που αφορά την Πολωνία όπου υπάρχουν χαμηλοί ε, μισθοί, χαμηλά έσοδα και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δοθούν ενισχύσεις για να προσαρμοστεί αυτό το πλαίσιο εργασίας. Κύριε Ανδρέσεν. κυρία Πρόεδρε. Το ίδιο ερώτημα όπως ο προλαλής σας είχα να θέσω κι εγώ. Και επανέρχομαι σε αυτή την κατάσταση. Στο μέλλον, εσείς στο μέλλον κυρία Αλμούνια, θα εγκρίνετε κρατικές επιδοτήσεις σε περιπτώσεις που γνωρίζετε ότι οι συνέπειες μιας τέτοιας πράξης θα απαιτήσουν να υπάρξει και κοινοτική αρρωγή. Σας ξαναλέω αυτό το οποίο είπα στον προηγούμενο ερωτώντα. Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των δύο αυτών των πραγμάτων. Εάν υπήρξε μια τέτοια σχέση, εγώ δεν θα μπορούσα να εγκρίνω μια κρατική επιδότηση η οποία βασίζεται σε επενδύσεις οι οποίες προκύπτουν από μια μετακίνηση η οποία κοστίζει χρήματα στον κοινωτικό προϋπολογισμό. Αλλά δεν υπήρξε κάποια τέτοια σύνδεση. Μα είναι σαφές, λέει κυρία Αντρίεσεν, όταν πήρατε την απόφαση Εγκρίνεται τη μετακίνηση ενός εργοστασίου από μια χώρα σε μια άλλη, ότι κάποιοι θα χάσουν τη θέση εργασίας τους. Δεν μπορείτε να αποκλείσετε λοιπόν κάτι τέτοιο όταν παίρνετε <clears throat> την απόφαση να εγκριθεί μια κρατική επιδότηση. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό έχει μια επίπτωση στο χώρο από τον οποίο θα μετακινηθεί το εργοστάσιο. Δεν μπορείτε να πείτε απλώς ότι είναι άσχετα τα δύο αυτά γεγονότα. Υπάρχει σαφής σύνδεση. Εάν υπάρχει μια κρατική βοήθεια για την εγκατάσταση ενός εργοστασίου, αυτό θα αναγκάσει, μάλλον θα ευνοήσει κάποιους να μετακινήσουν τα εργοστάσια τους σε αυτή τη χώρα και αυτό θα καταργήσει θέσει εργασία στι χώρε από τι οποίε έρχονται τα εργοστάσια. Δεν μπορείτε λοιπόν να τα αποσυνδέσετε. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Όταν εσεί αξιολογείτε μια κρατική επιδότηση σε αυτή την περίπτωση, θα έχετε στο μυαλό σα ότι αυτό θα κάνει αναγκαστική τη χρήση, την προσφυγή στο Ταμείο Παγκοσμιοποίηση για να καταπραγηθεί η κατάσταση για αυτού που χάνουν τη θέση εργασία του. Γενικά, λέει ο κ. Σαλμούνια. Δεν είναι παίγνιο μηδενικού αθρίσματος. Γενικά μια νέα επένδυση δημιουργεί νέα παραγωγή, νέα πλούτο, νέες θέσεις απασχόλησης. Μια νέα επένδυση δεν βασίζεται κατά ανάγκη στην κατάργηση προηγουμένων θέσεων απασχολήσεως και παραγωγή σε άλλο, σε άλλο Γιατί αλλιώς τελικά η συνολική ανάπτυξη θα ήταν μηδονική. Αυτό το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε είναι στην περίπτωση της ΔΕΛ, αν η ΔΕΛ της Ιρλανδίας και η ΔΕΛ της Πολωνίας, αν η επένδυση στην Πολωνία ήταν αποτέλεσμα του κλεισίματος του εργαστασίου στην ε, Ιρλανδία. Οι πληροφορίε που είχα σαν επίτροπο, όχι σαν αρμόδιο για κοινωνικά θέματα ή τον ανταγωνισμό, αυτά που έχω σαν πληροφορία είναι ότι δεν υπήρχε σύνδεση τη επένδυση με το κλείσιμο του εργοστασίου. Ευχαριστώ. Ο τελευταίο γύρο. Η κυρία Χούμπνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα κύριε Επιτροπέ. Από αυτά τα οποία μας είπατε βλέπουμε και επαγγελματισμό και αισιοδοξία και γνωρίζετε πως κληρονομήσατε στην Ευρώπη, στην τομέα της αρμοδιότητάς σας, ε, ένα βάρος ε, κρατικών ενισχύσεων και στις τράπεζες στο οποίο αναφερθήκατε αναλυτικά, αλλά και στην πραγματική οικονομία, στις βιομηχανίες και στις επιχειρήσεις. Και θα ήθελα να γίνετε κάπως πιο συγκεκριμένος για το πώς σκοπεύετε να προχωρήσετε για να αντιμετωπίσετε αυτή την πρόκληση όσον αφορά τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πραγματική οικονομία, όχι στον χρηματοοικονομικό τομέα. Τι γνωρίζει η Κομισιόν για την ομότητα των πρόσφατων αποφάσεων των κρατών μελών στο πλαίσιο της κρίσης. Και στην στρατηγική εξόδου από την κρίση, τι μπορείτε να κάνετε συγκεκριμένα για να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, των απαιτήσεων του Συμφώνου Σταθερότητας και της ανάγκης αναδιάρθρωσης, ε, απασχόλησης και του να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλάτε, μιλήσατε για μεγάλες κρατικές ενισχύσεις. Εάν δεν είναι λάθος τα νούμερα που έχω εγώ, εάν αφαιρέσουμε τις κρατικές ενισχύσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης που εγκρίθηκαν με το προσωρινό πλαίσιο που υιοθετήθηκε, ακριβώς λόγω της κρίσης, εάν τα αφαιρέσουμε αυτά, οι κανονικές ας πούμε κρατικές ενισχύσεις είναι γύρω στο 0,5% του ΑΕΠ της Ένωσης οπότε είναι χαμηλότερες από το επίπεδο που ήταν στην αρχή της δεκαετίας. Οπότε μόνο η κρίση οδήγησε στην αύξηση και το ερώτημα και συμφωνώ μαζί σας είναι πώς θα βγούμε από αυτό το προσωρινό πλαίσιο όταν υποχωρήσει η κρίση. Πότε και πώς. Και όπως ε, γίνεται και στην δημοσιονομική πολιτική και στην νομισματική πολιτική ε, υπάρχουν έκτακτα μέτρα σε καιρούς κρίσης. Η θέση μου είναι πως πρέπει να συζητήσουμε τώρα τη στρατηγική εξόδου πρέπει τώρα να ξεκαθαρίσουμε τι πρέπει να κάνουμε για να φύγουμε από το εξαιρετικό και προσωρινό αυτό πλαίσιο, το έκτακτο αυτό πλαίσιο, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πότε θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ακόμα δεν έχουμε ξεμπλέξει. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από ένα χρόνο, δεν είμαστε σε ελεύθερη πτώση. Βλέπουμε πως κάποια κράτη-μέλη είναι ξανά σε, ε, βρίσκονται σε θετική πορεία, το δικό στο κράτος μέλος όχι, αλλά είναι μεγάλος ο κίνδυνος και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τα, τη σταδιακή προσέγγιση. Εάν πάνε καλά τα πράγματα, και σύμφωνα με το σενάριο και την πρόβλεψη που έχουμε κάνει, το προσωρινό πλαίσιο για την μη το μη χρηματοοικονομικό κομμάτι θα τελειώσει το τέλος του 2010 και συγκεκριμένα για το για τα χρηματοοικονομικά έχει ξεκινήσει η συζήτηση σε επίπεδο κοφήν για το πότε. Αλλά δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε απόφαση. Πριν το τέλος του 2009 είπαμε πως δεν πρέπει να λάβουμε ακόμα την απόφαση, πρέπει να είμαστε σόφρονες. Στο μέλλον, όταν περάσουν όλα αυτά, πρέπει να εμβαθύνουμε αυτό το οποίο είχαμε ξεκινήσει πριν την κρίση και κατά τη διάρκεια της κρίσης, δηλαδή να υπάρξει οικονομική ανάλυση των κρατικών ενισχύσεων και να... Ναι, ναι, κυρία Πρόεδρε, να χρησιμοποιήσουμε βεβαίως την ανάλυση κόστους ωφέλους. Μπορείτε να επανέλθετε αν θέλετε. Δεν έχω ερώτηση. Μία πρόταση θα πω. Βεβαίως το 0,5% του ΑΕΠ είναι χαμηλό, αλλά είναι, κατανέμεται άνισα. Άλλα κράτη-μέλη δεν δώσαν τίποτα και άλλα δώσαν πολύ μεγάλο ποσοστό. Συμφωνώ πλήρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή η ανισοκατανομή του 0,5, αλλά όλα τα κράτη-μέλη, μεγάλα, μικρά, νέα, παλιά, οφείλουν να συμμορφώνονται με τον κανονισμό κρατικών ενισχύσεων. Ευχαριστώ παραμείναμε μέσα στον χρόνο. Η κυρία Ντάτη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, υποψήφιε Επίτροπε. Η κρίση που διατρέχουμε σήμερα μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε την νομοθεσία αλλά και την προσέγγιση που έχετε ακολουθήσει μέχρι στιγμή. Θέλω την άποψή σας για δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μία μπορεί να φαίνεται ίσον, η άλλη πολύ πιο σημαντική γιατί δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, αλλά τον κόσμο. Καταρχήν, η μεταρρύθμιση του κανονισμού για τα αυτοκίνητα που ενεκρίθη το Δεκέμβριο, που κατά την άποψή μου θέτει σε κίνδυνο την ελευθερία του επιχειρήν. Γιατί αυτό σημαίνει μείωση του αριθμού των εταιριών και την έλλειψη της δυνατότητας να πουλούν οι επιχειρήσεις την ε, επιχείρηση και τα εργοστάσια τους σε αυτόν τον οποίο επιλέγουν. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο λοιπόν είναι να υπάρξει μια τροποποίηση αυτού του κανονισμού γιατί βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης και αυτός ο, ο κανονισμός έχει να κάνει με πάνω από 300 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χιλιάδες θέσεις εργασιών. Παρά τις ε, δηλώσεις του <clears throat> Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για τα θέματα αυτά για τον φόρο άνθρακος στα ευρωπαϊκά σύνορα, παρά το γεγονό ότι δεν υπήρξε επιτυχία στην Κοπεχάγη, μήπω αυτά πρέπει να σα αναγκάσουν να ξανασκεφτείτε για ένα φόρο άνθρακο στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι απαραίτητο η Ευρώπη να προστατεύσει τι επιχειρήσει τη από τον αθέμητο ανταγωνισμό χωρών όπου δεν υπάρχουν καθόλου περιορισμοί που να προστατεύουν το περιβάλλον. Και παρέχομαι σε αυτά που είπε ο πράσινο, ο συνάδελφό μου από του πράσινου, ότι πρέπει τελικά η προστασία του περιβάλλοντο να είναι παράγον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ για τους κανονισμούς σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, όπως ξέρετε, υπήρξε μια μακρά διαδικασία διαβούλευσης, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμμετάσχει πλήρως. Η Κομισιόν δεν έπαιξε ρόλο μονάχα σε αυτή τη διαβούλευση, αλλά εξέδωσε μια ανακοίνωση, παρουσίασε ένα σχέδιο κανονισμού. Ελπίζουμε να περατώσουμε τις διαβουλεύσεις και να εγκρίνουμε τον νέο αυτό κανονισμό το Μάιο ή προηγουμένως. Τι λέει λοιπόν αυτό το σχέδιο κανονισμού. Διατηρούμε κάποιες παρεκκλήσεις από το γενικό κανονισμό ανακατηγορία σε ό,τι αφορά τις επισκευές στις ε, επισκευές λοιπόν των αυτοκίνητων και σε ό,τι αφορά τα ανταλλακτικά. Και θα προτείνουμε να υπάρξει συμπερίληψη στο γενικό καθεστώς των ε, διανομέων, των αντιπροσωπιών των αυτοκινήτων. Εμείς προσπαθήσαμε να προωθήσουμε μια πολυμαρκική μορφή αντιπροσωπιών, δηλαδή αντιπροσωπίες να εκπροσωπούν πολλές εταιρείες και να μην υπάρχει μονάχα το να μην υπάρχει μονάχα αντιπρόσωπο για μια εταιρεία να υπάρχει δυνατότητα πραγματικού ανταγωνισμού στο επίπεδο των ε, αντιπροσωπιών. Εγώ δεν διακρίνω τον κίνδυνο τον οποίο αναφέρατε εσείς, αλλά εγώ είμαι ανοιχτό για να εξετάσω το θέμα αυτό μέσα στη διαδικασία αυτή συζητήσεων και διαβουλεύσεων τα προβλήματα αυτά τα οποία θα πρέπει να επιλύθουν μέχρι το Μάιο. Έχουμε το χρόνο να τα εξετάσουμε αυτά. Για το θέμα του φόρου άνθρακος, εγώ δεν είμαι δεν είμαι εμπειρογνώμων. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς το ίδιο θέμα το οποίο έθεσε ο κύριος Γκίγκολτ και ο κύριος Λάμπερτς. Ο φόρος άνθρακος στα σύνορα είναι κάτι που προτιμώ να μην το συζητήσω γιατί πιστεύω ότι θα καταλήξουμε μετά την Κοπεχάγη σε κάποια λύση. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής χωρίς να χρησιμοποιήσουμε προστατευτικού χαρακτήρα εργαλεία, γιατί τότε θα χάσουμε όχι μόνο στα θέματα του περιβάλλοντος, αλλά και σε εμπορικό και οικονομικό επίπεδο. Σύντομη ερώτηση, συμπληρωματική αν θέλετε, για το τελευταίο θέμα. Εγώ επανέρχομαι σε αυτά που έλεγε η κυρία Γκούλαρτ πώς θα εξηγήσετε στους Ευρωπαίους πολίτες και φορολογούμενους και μισθωτούς ότι οι, επιχειρήσει του επιχειρήσεις τους προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά αυτό είναι σε βάρος της θέσης εργασίας τους. Γιατί άλλες παγκόσμιες επιχειρήσεις δεν προστατεύουν το περιβάλλον και αυτός είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποια παιδαγωγική εργασία για να καταλαβαίνουν και οι εργαζόμενοι γιατί χάνουν τις θέσεις απασχόλησής τους προς όφελος επιχειρήσεων που δεν σέβονται το περιβάλλον. Επιμένω, σας λέω ότι δεν ήταν ακριβώς το ίδιο σημείο. Σίγουρα θα πρέπει η Ευρώπη να επεξεργαστεί αυτό το θέμα και η Ευρώπη έχει μια πολύ καλή αφετηρία για να μπορέσει να εργαστεί τους επόμενους μήνες για μια συμφωνία για τα κλιματικά θέματα που να επιλύσετε τα προβλήματα τα οποία αναφέρετε. Είναι πραγματικά προβλήματα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια όταν υπάρχουν αναδυόμενες χώρες οι οποίες είναι πολύ ανταγωνιστικές λόγω τους χαμηλού μισθολογικού επίπεδου και συγχρόνως δεν έχουν αναλάβει κανένα, καμία δέσμευση για να αγωνιστούν κατά της κλιματικής αλλαγής. Αλλά δεν είναι το μόνο σενάριο. Το πραγματικό σενάριο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε είναι η επίτευξη μια συμφωνία και πρέπει να κάνουμε μεγάλε προσπάθειε. Είδαμε στην Κοπεχάγη πόσο δύσκολο είναι να φτάσουμε σε μια τέτοια συμφωνία. Είδαμε όμω στην Κοπεχάγη ότι αν η Ευρώπη δεν παίξει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία αυτή δεν θα υπάρξει συμφωνία. Η ευθύνη μας λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Δεν τίθεται μονάχα θέμα συμφέροντος, τίθεται και θέμα ευθύνης για την κλιματική αλλαγή. Ενώπιον της κλιματικής αλλαγής μάλλον. Ο κύριος Κάζα έχει το λόγο. θα επανέλθω σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και όπως αναφέρθηκε σε καιρούς χρηματοπιστωτικής ε, κρίσης υπάρχει ε, στρέβλωση του ανταγωνισμού εξαιτία των κρατικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις. Είσαστε ικανοποιημένος από τις, πολιτικές, τις ισχύουσες πολιτικές και θα είχατε κάνει κάτι διαφορετικά αν έπρεπε να αποφασίσετε τώρα. Θυμάμαι ότι όταν συζητήσαμε την εισδοχή της Ισλοβακίας και της Μάλτας στην Ευρωζώνη, είπατε ότι ο προστατευτισμός οδηγεί στην στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Το πιστεύετε ακόμα κύριε υποψήφιε. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως κύριε Κάσα. Πιστεύω σε αυτή την αρχή. Η κρατική ενίσχυση είναι και καλή και κακή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δημόσιο χρήμα για να αντιμετωπίσουμε τις αποτυχίες της αγοράς ή να ενθαρρύνουμε ορισμένες πολιτικές ε, που είναι ελληματικές από τους μηχανισμούς της αγοράς ή που οδηγούν σε άδικη κατανομή και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δημόσιο χρήμα για να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις δραστηριότητες. Πολιτικά μπορούμε να το συζητήσουμε ποιο είναι το επίπεδο αποδοχής, που είναι τα όρια, τι είναι πιο αποδοτικό. Αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική συζήτηση, αλλά το γεγονό ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το δημόσιο χρήμα για καλούς σκοπούς, αυτό είναι ε, αμετακίνητη πεποίθησή μου παράλληλα γνωρίζω ότι δεν χρησιμοποιούμε πάντα το δημόσιο χρήμα προς ε, έναν καλό σκοπό για ένα καλό σκοπό. Άρα ε, οι κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το, το πλαίσιο, θα πρέπει να βελτιωθούν οι κρατικές ενισχύσεις όπως έγινε και πριν από την κρίση. Τώρα αντιμετωπίσουμε τις απόρριες της κρίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα έκτακτο, μια έκτακτη πλαισίωση και μετά θα συνεχίσουμε με την προσαρμογή. Γι' αυτό προετοιμάζουμε και την αξιολόγηση των, της αποδοτικότητας των κρατικών ενισχύσεων. Το 2005 είχαμε το πρόγραμμα δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Είχαμε μία ε, οικονομική προσέγγιση, μαθαίνουμε από την πείρα και τα λάθη μας, αλλά νομίζω ότι πάντα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι η καλή χρήση του δημόσιου χρήματος θα πρέπει να ελέγχεται πάντα ε, χρησιμοποιώντας ε, ή μάλλον με βάση την κακή χρήση του δημοσίου χρήματος πολλές φορές. Και πολλές φορές οι κυβερνήσεις χρειάζονται πόρους που πρέπει να χρησιμοποιήσουν. Βρισκόμαστε σε μια εσωτερική αγορά και μας ενδιαφέρει και η συνοχή. Γι' αυτό στις εξαιρέσεις από κρατικές ενισχύσεις λαμβάνουμε υπόψη πολλές φορές στον περιφερειακό παράγοντα. Συμφωνώ ότι θα υπάρξει στρέβλωση της, στην εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό καθεαυτό. Πιστεύω όμως παράλληλα ότι θα πρέπει να έχουμε μία βιώσιμη στρατηγική διεξόδου. Δεν πιστεύετε ότι με όλες, με όλες αυτές τις στρεβλώσεις θα πρέπει να αποφασίσουμε πότε θα αποχωρήσουμε από αυτό το πλαίσιο, πότε θα έχουμε μια τέτοια στρατηγική εξόδου γιατί μιλήσατε για το ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά προείπατε ότι είναι πολύ πρόημο να αποφασίσουμε για αυτή τη στρατηγική εξόδου. Εγώ νομίζω ότι είναι επίγον το ζήτημα. Θα πρέπει να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εξέλθουμε από αυτό το πλαίσιο απάντηση. Εάν διαβάσετε προσεκτικά ε, αυτά που προείπα, θα δείτε μία απόχρωση στον τομέα των, του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δεν ανέφερα, δεν αναφέρθηκα σε μία ημερομηνία. Ως προς το μη χρηματοπιστωτικό τομέα, το μη χρηματοδοτικό πλαίσιο, μίλησα ε, για το 2010, το Δεκέμβριο του 2010. Αυτή είναι η προθεσμία. Καταρχήν, θα ήθελα να, θέλω να πιστεύω ότι θα έχει λήξει η κρίση μέχρι τα τέλη του 2010 και θα μπορώ να το κάνω αυτό, αλλά υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Ευχαριστώ, περνάμε στον κύριο Φέρμπερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Αλμούνια. Ήδη σήμερα συζητήσαμε τα της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αναφερθώ και εγώ σε αυτά τα οποία είπε η κυρία Ντατή Έχουμε μια σειρά μεταρρυθμίσεων ε, φέτος που είναι στην ημερήσια διάταξη όσον αφορά κάποια ζητήματα. Θα ήθελα να σα ρωτήσω πώς τοποθετήσετε σε αυτό σχέση με τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε ότι έχω γραπτό έργο ε, δεν χρειάζεται να σας πείσω ότι θα πρέπει να υπάρχει αγαστή σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον. Σας έχω πείσει εδώ και 5,5 χρόνια γι' αυτό, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων μου. Κάθε φορά που θελήσατε, ε, προσήλθαμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ όταν θελήσατε να το συζητήσουμε στην Ολομέλεια, το συζητήσαμε και με τους συντονιστές και με τα μέλη της ε, Επιτροπής. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με την ε, ε, πρόεδρο της ΕΚΟΝ, όπως και με την κυρία Μπόουλς τώρα. Όταν μιλάμε για ανταλλαγή απόψεων, εγώ είμαι πάντα διαθέσιμος και στις, και στις αποφάσεις που θα λάβω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι κοινωνός. Σε περίπτωση τακτικής διαδικασίας θα ε, ακολουθήσω αυτή την πλαισίωση. Θα δούμε πώς θα έχουν οι μελλοντικές ρυθμίσεις ως προς τις συλλογικές αποζημιώσεις. Στο τομέα του ανταγωνισμού υπάρχουν πολλές αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή αφεαυτής. Δεν θέλω να σας πω τώρα πώς θα λάβω αυτές τις αποφάσεις. Δεν μπορώ να το προδικάσω όπως ισχύει για την αυτοκινητοβιομηχανία. Γίνεται ανοιχτή διαβούλευση μέχρι τέλους και όσον αφορά την εφαρμογή ε, μέτρων ανταγωνιστικότητας που αφορούν ζητήματα εμπιστευτικού χαρακτήρα. Μπορώ να σας πω εξ post τι απόφαση θα έχουμε λάβει και γιατί. Ευχαριστώ. Είναι καλό το ότι θέλετε να έρχεστε εδώ πέρα. Αυτό το οποίο με αφορά εμένα για το block exemption είναι πως ε, η Κομισιόν θα διαγράψει το, το δίκαιο το οποίο μετά θα εφαρμόσει χωρίς να ακούσει και κανέναν. Οπότε το ερώτημα είναι Έχουμε και εμπειρία με προκατόχους σας ε, και το ερώτημα είναι αν θα συνεργαστείτε ε, τόσο στενά όσο ο κύριος Κάρελ Φανμίρτ ε, ή η κυρία Κρούς. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε μεταξύ Φανμίρτ και Κρούς εσείς που θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας. Νομίζω ότι στο, ε, θα πρέπει να επιλύσουμε αυτά τα ζητήματα στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, κάτι το οποίο θα προσπαθήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω κύριε Επίτροπε και εγώ με τη σειρά μου έχετε μεγάλη πείρα και υπάρχουν πολύ υψηλές προσδοκίες. Θα ήθελα να αποβάλω δύο ερωτήσεις. Με βάση τα μέσα που διαθέτεται θα, θα υπάρχει καλύτερη προσβασιμότητα ως προς την πίστοση για τις επιχειρήσεις. Τι θα κάνετε στον τομέα του ανταγωνισμού για να μην πληγούν οι ΜΜΕ ως προς τις κρατικές ενισχύσεις. Όταν βγούμε από αυτή την έκτακτη συγκυρία θα έχουμε ε, διάφορες παρεμβάσεις. Το 85% των κρατικών ενισχύσεων ε, αφορούσε ε, μία συγκεκριμένη στοχοθέτηση. Αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι τις τομεακές έρευνες και δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να μας απασχολήσει και η διανομή των ε, τροφίμων ή ε, προϊόντων της διατροφικής ε, αλυσίδας που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στον τοπικό, στον εγχώριο τομέα. Σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό και την πρόσβαση στις πιστώσεις, πώς θα υπάρχει ροή πιστώσεων στις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ, που δεν έχουν τόσο μεγάλη πρόσβαση στις κεφάλαια αγορές. Βεβαίως, με σχέδια αναδιάρθρωσης μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Έτσι ώστε αυτοί που δεν αποδίδουν τόσο καλά για να παραμείνουν στην αγορά δεν θα μπορούν να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να στρεβλώνουν ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα ή το χρηματοπιστωτικό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την φερεγγιότητά τους, τους ισολογισμούς τους, διαφορετικά δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πιστώσεις, διότι χρειαζόμαστε την εξυγίανση του τομέα, την επανακεφαλαιοποίηση, το, έναν σωστό ισολογισμό, κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο την πολιτική ανταγωνισμό, αλλά και τις κρατικές ενισχύσεις. Ως προς τις ε, τομεακές μελέτες αποτελούν ένα πολύ ισχυρό μέσο. Κατά την προηγούμενη θητεία θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο μελέτες στον τομέα της ενέργειας και στον τομέα των φαρμακευτικών σκευασμάτων που θα μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία έτσι ώστε να ενισχύσουμε μία πολιτική ανταγωνισμού. Υπάρχουν πολλά προβλήματα ανταγωνισμού και εάν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα ε, προβλήματα από ευρωπαϊκή σκοπιά ή εθνική σκοπιά, θα το δούμε αυτό για να δούμε ποια είναι η πιο επιτυχής ε, προσέγγιση. Δευτερολογώντας, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ε, με βάση τις φιλοδοξίες σας, πώς βλέπετε την ευρωστία του, του σώματος έτσι ώστε να έχετε τα ε, σωστά χρηματοδοτικά μέσα ή επιπρόσθετα ε, μέσα στήριξης. Πιστεύετε ότι αυτό παραμένει πρόβλημα ή έχει επιληθεί. Ο μελλοντικός ε, γενικός διευθυντής και άλλοι υπεύθυνοι θα χαίρονταν να σας δώσουν μία απάντηση. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με, εξαιρετικές, με μια εξαιρετική υπηρεσία. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Από το 2004 ε, διευρύνουμε τις αρμοδιότητές μας με νέες προτεραιότητες, αλλά δεν μπορώ να σας πω από την πρώτη μέρα ότι δεν χρειάζομαι επιπρόσθετα μέσα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα μέσα που διαθέτουμε, αλλά τώρα, εάν στο μέλλον κρίνω ότι πρέπει να επεκταθούν και δεν μπορούμε να επιτελέσουμε αυτό το έργο με, τους, με το προσωπικό των χιλίων ατόμων, θα ζητήσω ε, επιπρόσθετη στήριξη. Ευχαριστώ. Ο το ζήτημα των προστήμων σε περιπτώσεις παραβιάσης των κανόνων του ανταγωνισμού, ιδίω από καρτέλ, έχει διαδραματίσει ήδη στο παρελθόν ένα σημαντικό ρόλο. Αλλά πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό, κύριε Αλμούνια, και να δούμε μια ιδιαίτερη πλευρά του. Η Κομισιόν δεν πρέπει να παρετηθεί της ε, δυνατότητος να δράσει εκεί. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση και δίωξη των παραβιάσεων των καρτέλ και δεν πρέπει να αφήσει τα πράγματα να συνεχίσουν έτσι. Τίθεται όμως το θέμα της διαφάνειας. Μπορείτε εσείς να φανταστείτε να υπάρχουν κάποια, ένας κατάλογος κριτηρίων για το πότε επιβάλλονται κυρώσεις και σε ποιο επίπεδο που να, μπορούμε να, να μπορείτε να τις συζητήσετε με το Κοινοβούλιο γιατί δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος κατάλογος μέχρι τώρα πολλές φορές έχει χάσει σε αγωγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η Κομισιόν γιατί δεν υπήρχε και ιδιαίτερη διαφάνεια σε σχέση με την επιβολή προτάσεων. Μήπως θεωρείτε ότι χρειάζεται ένας περαιτέρω διάλογος για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα των κυρώσεων και πάντα είμαι ανοιχτός στη συζήτηση αυτού του θέματος. Θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα των κυρώσεων μέσα στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής ανταγωνισμού. Υπάρχουν όμως γνωστά κριτήρια, υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν το 2006 για τις κυρώσεις που επικαιροποιούν την συσσωρευμένη πείρα μας από την θέση σε ισχύ του κανονισμού που αποτελεί την νομική βάση για τις κοινώσεις. Είναι ο κανονισμός 1 κάθετος 2003, αν θυμάμαι καλά. Αναφερθήκατε στις αποφάσεις του ΔΕΚ που πάντα τηρούμε και σεβόμαστε αλλά θα ήθελα να σας ε, θέσω ένα παράδειγμα κυρώσεων που εγκρίθηκαν μετά από τις κατευθυντήριες γραμμές του 2006 που διορθώθηκαν από το ΔΕΚ. Και από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να μας καταδεικνύει ότι το, το ΔΕΚ θα λάβει αποφάσεις που να αντιτίθενται σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη. Αυτό μπορεί να το συζητήσουμε. Αν μετά από το 2006 τα πράγματα είναι ακριβώς όπως το λέτε. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι έτσι. Εγώ θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία λαμβάνονται οι συγκεκριμένες αποφάσεις και πώς γίνεται κάτι το οποίο δεν είναι στη διακριτική ευκαιρία του αρμόδιου επιτρόπου ή της αρμόδιας επιτρόπου. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει διευκρίνηση εκεί. Δεύτερον, εσείς μπορείτε να σκεφτείτε με τέτοιες ε, κυρώσεις, τις οποίες εγώ δεν τις απορρίπτω, όταν υπάρχουν θέσεις εργασίες οι οποίες διακυβεύονται, θα μπορούσατε να φανταστείτε αυτά τα κριτήρια να περιλαμβάνουν και κοινωνικές ρήτρε σε ό,τι αφορά την προστασία των θέσεων απασχόλησης. Και αυτό ίσως θα πρέπει να τεθεί σε δημόσια συζήτηση. Δεν πιστεύω ότι είναι σαφές αυτό σε επαρκές επίπεδο ενώπιον της κοινή γνώμης ότι λαμβάνει υπόψη αυτό το κριτήριο. Ειλικρινά νομίζω ότι επεξηγούνται επαρκώς στις κατευθυντήριες γραμμές με βάση τον αντίστοιχο κανονισμό που προϋπήρχε, δηλαδή οι κυρώσεις υπολογίζονται ανάλογα με την δημιουργηθήσα ζημία από την κατάχρηση των αρχών ανταγωνισμού. Επίσης θα αυξάνονται ανάλογα με την βαρύτητα της ζημίας που δημιουργείται, όχι μόνο του μεγέθους, αλλά και της σημασίας, του βάρους και ανάλογα με το χρόνο που ίσχυσε η, πολιτική κατά του ανταγωνισμού. Πρόκειται για πολύ σοβαρά κριτήρια τα οποία την χάνουν υποστήριξης. Υπάρχει όμως ε, και μια δυνατότητα που είναι η εξή. Εάν μια επιχείρηση που αποτελεί αντικείμενο κύρωσης ισχυριστεί με επαρκή επιχείρηματα ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην κύρωση, στην χρηματική αυτή κύρωση, μπορεί να υπάρξει μια διαφοροποίηση στην καταβολή της ε, κύρωσης, το ability to pay που εφήρμοσε Επιτροπή στις ε, εξάντε κατευθυντήριες αγαραμές που χρησιμοποιήσετε, δηλαδή όταν δεν υπάρχει δυνατότητα καταβολής ε, του προστίμου. Θα πρέπει βεβαίως να γνωρίζουμε κατά πόσο η ε, Επιτροπή μετατρέπει την κατάστασή της έτσι ώστε να μην καταβάλει το πρόστιμο θα πρέπει να δούμε κατά πόσο βρίσκεται σε αντικειμενική δυσχέρεια να καταβάλει αυτό το πρόστιμο. Δηλαδή, εάν ε, τίθενται σε κίνδυνο οι θέσεις εργασίας, τότε θα υπάρχουν άλλα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από μία πολιτική ανταγωνισμού να αντιμετωπίσει όλες ε, τις ζημίες ε, που προκλήθηκαν από μία επιχείρηση και μόνο. Ωραία, σας ευχαριστούμε. Τελευταίος, αλλά οπωσδήποτε όχι έσχατος, ε, για τους φιλελεύθερους ο κύριος Τρεμόζα. Για δεύτερη φορά, σε δεύτερη ακρόαση, παίρνετε τελευταίο τον λόγο. Καλό απόγευμα κύριε Ελμούνιο, δείξατε μεγάλη φαινεγιότητα ω ε, επίτροπο και όπω τα καλά κρασιά παλιώνοντα, βελτιώνεστε. Ω επίτροπο ε, ανταγωνισμού ξέρετε ότι η Ισπανία έχει πολλά, πολλούς φακέλους ανοιχτού στα θέματα ανταγωνισμού για λεγόμενες παράνομες κρατικές ενισχύσεις. Αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν περίπου 400 ανοιχτοί φάκελοι για υποτιθέμενες παράνομες ενισχύσεις του Ισπανικού κράτους σε διάφορους παραγωγικούς τομείς. Ξέρετε ότι η Ισπανία έχει ένα σημαντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΦΡΟΠΟ, το οποίο είναι το σχέδιο για την εξηγήση του τραπεζικού τομέα και επίσης διάφορα εργαλεία οικονομικής <clears throat> ενίσχυσης και πρόθεσης. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ε, ρυθμίσεις όπως αυτή για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δύσκολη θέση που ουσιαστικά οδηγούν σε τελμάτωση τη οικονομική δραστηριότητα. Εσείς κύριε Επίτροπε, όταν συγκρούεται το ευρωπαϊκό συμφέρον με το ισπανικό συμφέρον, πώς θα κινηθείτε. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> Και η, τα καλά κρασιά και τα κρασιά της Ριόχα και τα κρασιά της δικής σας περιοχής βελτιώνται πράγματι με το χρόνο. Η εθνικές βοήθειες ενισχύσεις της Ισπανίας είναι ίδιες με αυτές της Ελλάδος, της Λετωνίας, οποιασδήποτε άλλη χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μένα, μέσα στην άσκηση του καθήκον μου ως Επιτρόπου ε, Οικονομικών Θεμάτων ή ε, Ανταγωνισμού, το καθήκον μου είναι να εφαρμόσω τους ευρωπαϊκούς κανόνες, να σεβαστώ τις συνθήκες, να εφαρμόσω λοιπόν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το να ακολουθήσω την γενική πολιτική της Κομισιόν αυτό κάνω και αυτό το οποίο εγώ έχω υποσχεθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αυτό θα συνεχίσω να κάνω πάντα. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, κύριε Επίτροπε. Το, αεροδρόμιο της Βαρκελός δεν μπορεί να κάνει πτήσεις προς 23 χώρες γιατί υπάρχουν διμερείς συμφωνίες του Ισπανικού κράτους που το εμποδίζουν να κάνει κάτι τέτοιο και επιτρέπουν τέτοιες πτήσεις μόνο από το αεροδρόμιο της ε, ε, Μαδρίτης. Αυτό μπορείτε να το δείτε ότι πράγματι ισχύει. Πώς θα δράσετε εναντί αυτής της χτυπητής διάκρισης σε ανταγωνισμό. Όπως ξέρετε, στη Νέα Κομισιόν, οι κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των μεταφορών είναι αρμοδιότητες του Επιτρόπου Ανταγωνισμού. Εκεί λοιπόν που υπάρχει μια μη ανταγωνιστική αντιμετώπιση, μια παραβίαση κατά του άρθρου 101-102 των συνδικών, εγώ θα δράσω. Εγώ έχω θέσει μια γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν ακριβώς για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τα είδαμε αυτά τα ζητήματα αφού έφυγε η Επιτροπή Μεταφορών. Μην πείτε. Λοιπόν, τελείωσαν εδώ οι ερωτήσεις. Ο υποψήφιος κύριος Επιτροπός τώρα έχει πέντε λεπτά να συνοψίσει και ίσως έχει ήδη λάβει το, το έγγραφό μου. Έχω σημειώσει πως έχετε υποσχεθεί στον κύριο Φέρεμπερ πως θα είστε καλύτερος από τους καλύτερους. που νομίζω είναι το ίδιο με αυτό το οποίο αναφέρεται στο σημείο 1, με το νούμερο 1. Τέλος πάντων, θα ήθελα και εγώ να ακουστεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς, αλλά είδα al προφανώς τα τρία αυτά σημεία που αναγνώσατε στην αρχή και τα οποία μου έδωσε ο γραμματέας της Επιτροπής, σας συμφωνώ απόλυτα. Δεν ξέρω αν πρέπει να υπογράψω ενώπιον των βουλευτών και να δηλώσω δημόσια ότι συμφωνώ με αυτά τα οποία ζητείτε για τα θέματα της πληροφόρησης. Εγώ συμφωνώ και σας λέω και πάλι ότι θα σας διατηρώ ενήμερους στα θέματα αυτά που είναι μεταξύ χαρτοφυλακίων και επίσης σας <laughs> δίνω το έγγραφο αυτό υπογεγραμμένο για αυτά που λέτε στην τρίτη παράγραφο Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Όχι γιατί μου δώσατε κάτι να υπογράψω, αλλά για την ανταλλαγή απόψεων και όλες τις ερωτήσεις που θέσατε, όπως είπα προηγουμένως. Ελπίζω ότι αυτό θα είναι και ο κανόνας σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας, να υπάρχει πραγματικά μια ανταλλαγή απόψεων σε βάθος για όλα τα θέματα τα οποία άπτονται τη πολιτική αυτής ανταγωνισμού, που θεωρώ πάντα ότι είναι πάρα πολύ κεφαλαιόδης για τη λειτουργία της εσωτερική αγορά και της ευρωπαϊκής ε, αγοράς. Προτού αναλάβω αυτό το λειτουργήμα, επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή. Δεν είναι ένα πολιτικό λειτουργήμα που έχει να κάνει με μια προσωπική <clears throat> αντιμετώπιση ή άποψη. Είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την ευρωπαϊκή πεποίθησή μου ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί να γίνεται το έργο αυτού της, του ελέγχου του ανταγωνισμού προς όφελος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και οι προσπάθειες που έχουν γίνει πολλές φορές δύσκολες προσπάθειες έχουν βοηθήσει χώρες μας να ξεπεράσουν πολλές δυσκολίες. Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι έχουμε καταφέρει πολλά θετικά σε επίπεδο Ευρώπης. Πάντα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις και θα συνεχίσει αυτό να ισχύει για τα επόμενα χρόνια. Και στη δική μου περίπτωση, εγώ έχω συμμετάσχει με υπό την προηγούμενη ιδιότητά μου σε πολλές συνεδριάσεις των G20 για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και να δούμε τι κόσμος, πώς θα είναι οργανωμένος ο κόσμος στην, στις αρχές του 21ου αιώνα, πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση και είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ότι έχουμε ένα πολύ δύσκολο και σημαντικό έργο και η Κομισιόν και εσείς ως Κοινοβούλιο που έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα η θέση σας από την Συνθήκη της Λισαβόνας και εξάλλου και το Συμβούλιο το οποίο μερικές φορές δεν φαίνεται να έχει την ίδια φιλοδοξία σαν θεσμός και την ίδια ορμή ευρωπαϊστικού χαρακτήρα όπως έχουν τα, ευρωπαϊκά, τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά νομίζω ότι η συνεργασία των τριών αυτών θεσμικών οργάνων θα εξέλθει μια Ευρώπη ενισχυμένη και της οποίας ο ρόλος θα αναγνωριστεί από τους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Μέχρι και στην ώρα μας τελειώσαμε. Να σας υπενθυμίσω πως η ακρόαση αξιολόγηση είναι 8 η ώρα, 1G3 σε μισή ώρα. 8 η ώρα. Και εγώ είμαι κουρασμένη.